Euh, Καλημέρα σας. Με πολύ μεγάλη χαρά συμπροεδρεύω της ακρόασης αυτής. Όπως ξέρετε, φαντάζομαι, πρόκειται για ένα μείζον ζήτημα, το οποίο και εγώ εργάζομαι εδώ και 20 χρόνια. Με χαρά λοιπόν να βλέπω σήμερα τα ζητήματα των, παράνομων, των όρων παράνομων χρημάτων, το θέμα της διαφθοράς και του πώς αυτή επηρεάζει τις αναπτυσσόμενες χώρες να είναι στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για ένα δολάριο βοήθειας αναπτυξιακής, οι φτωχές χώρες χάνουν 10 δολάρια σε παράνομες οικονομικές ροές. Αυτό οφείλεται Μάλλον αυτό προέρχεται σε πολλές, από πολλές έρευνες που δείχνουν ότι οι παράνομες αυτές ροές είναι ουσιαστικά το δεκαπλάσιο της αναπτυξιακής βοήθειας. Πρόκειται για τροχοπέδι στην ανάπτυξη και στην δυνατότητα των χωρών να παράσχουν τις βασικές ε, κοινοφελείς υπηρεσίες πολίτες. Και ενώ οι κυβερνήσεις περιορίζουν σημαντικά τις ενισχύσεις τους, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύο μάστιγες που οδηγούν σε απώλειες δις για τις ανεψόμενες χώρες. Αυτό αποτελεί ανάγκη και μάλιστα κατεπίγουσα. Είναι σχεδόν τοπικό να υποστηρίζει κανείς αύξηση της αναπτυξιακής βοήθειας, εθελοτυφλώντας και μη βλέποντας τις επιχειρήσεις των πολυεθνικών και των άλλων φορέων και παραγόντων που με τη χρήση φορολογικών παραδείσων και τεχνικών φορολογικής βελτιστοποίησης στερούν ε, τα θεμητά ε, εισοδήματα από τις αντισώμενες χώρες. Αν παρά την κρίση οι Ευρωπαίοι συμπολίτε μας εξακολουθούν μασικά να στηρίζουν τη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια, θέλουν επίσης αυτή να είναι αποτελεσματική προς όφελος του πληθυσμού. Τα πολέμηση της διαφθοράς για μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρήση των ε, πόρων Παναπατρισμός ε, των παράνομης προέλευσης πόρων στις χώρες ε, προέλευσης, τα, τα αυτά χρήματα προέρχονται από πολυεθνικές είτε από οπουδήποτε, είτε από ε, αδίστακτους άλλους ηθήνοντες, ε, είναι κάτι το απαραίτητο. Αυτή την εποχή Είμαι στην ομάδα ΜΕΚ, που είναι μια αφγανική ε, οργάνωση, ε, μεικτή, δηλαδή αποτελείται και από Αφγανούς και από αλλοδαπούς και στόχο έχει την καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλήματος μαύρου χρήματος στο Αφγανιστάν. Έχουμε κάνει και την έκθεση αυτή που σας είχα πει χθε γιατί το σκάνδαλο με την ε, τράπεζα Καμπούλ Μπάνκ ήμουν στο Αφγανιστάν τις δύο τελευταίες εβδομάδες όταν και υπήρξε η απόφαση του δικαστηρίου για την υπεξαίρεση των 900 αυτών ε, εκατομμυρίων ε, ευρώ, ε, συγγνώμη, δολαρίων, τα οποία ουσιαστικά εκλάπησαν από τους ε, διευθύνοντες της τράπεζας και από ανθρώπους προσκύμενους στην κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Μπορείτε να διαβάσετε την ιστορία της απάτης αυτής στο blog που έχω ή αν πάτε και στο site της ε, οργάνωσης ΜΕΚ στο Αφγανιστάν. Το σκάνδαλο ποιο ήταν η απόφαση, η τιμιγορία. Δεν χρησιμοποιεί τους νόμους περί ε, ξέπλυματος δρόμικος χρήματος, επομένως δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια κατάσχεση, κάποια ε, δίμευση περισσιακών στοιχείων. Άρα αυτά τα 900 εκατομμύρια δεν μπορούν να ανακτηθούν. Βλέπουμε λοιπόν ε, ποια είναι η μεγάλη πρόκληση με τη σωστή εφαρμογή των κανόνων, των διεθνών κανόνων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ποια είναι τα αποτελέσματα της διαφθοράς. Με πάρα πολύ ενδιαφέρον θα ακούσω την παρουσίαση του κυρίου Πάρτο για αυτό το ζήτημα, για το Αφγανιστάν. Όχι βέβαια μόνο την παρουσίαση του κύριου Πάρτο, αλλά όλες τις παρεμβάσεις. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ταβάρης. Σας ευχαριστώ αγαπητή Εύα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω εδώ δύο επιτροπές, ε, την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή ΚΡΙΜ, την Ειδική Επιτροπή. Ουσιαστικά εμείς βλέπουμε την κρυφή πλευρά της κρίσης, την ε, εγκληματικότητα, αλλά πρέπει να δούμε και τη ροή ε, χρήματος που έχει προέλθει από ξέπλυμα από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κάποιε φορέ μάλιστα βοηθούν και τα νομικά και τα τραπεζικά συστήματα των, των αναπτυγμένων χωρών. Άρα δεν μιλάμε μόνο για κρίση στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ε, μιλάμε για μια παρέμβαση ουσιαστικά δόλια ε, στις ε, παγκόσμιες υποθέσεις και θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά με αυτό το θέμα. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε άλλο γιατί είναι πολλοί οι ομιλητές μας, πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις που θα ακούσουμε με τον ε, κύριο Raymond Baker, διευθυντή του Global Financial Integrity, που θα μας μιλήσει για το παγκόσμιο σκιώδες χρηματοοικονομικό σύστημα, για τα παράνομα χρήματα. Ο κύριος Βίμινγκ, που θα ήταν ο δεύτερος ομιλητής, είναι ένας ε, ανώτατος σύμβουλος της Βρετανικής κυβέρνησης ε, και θα μας μιλήσει για την ε, ποινικοποίηση του παράνομου χρηματισμού και το ρόλο του στην καταπολέμηση της διαφθοράς και μετά θα μας μιλήσει και η κυρία Τζένιφερ Πράμπλετ που είναι από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών κατά του ξεπλήματος. Αυτές είναι οι τρεις παρεμβάσεις. Θα δώσω στον κάθε μιλητή 15 λεπτά χρόνο. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρώτο κλάστερ, αυτή την πρώτη δέσμη, το πρώτο πάνελ και μετά θα ακούσουμε ε, και τους υπόλοιπους συναδέλφους που θα θέλουν το λόγο. Ας ξεκινήσουμε αντί για δεύτερο με πρώτο τον κύριο Βίνινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη των δύο επιτροπών που με κάλεσαν. Το θέμα έχει λησμονηθεί στη Δυτική Ευρώπη. Βλέπετε την πρώτη διαφάνεια. Ανεξήγητος πλούτος στην δημόσια διοίκηση. Παρέθεσα το άθρο 20 της συμβάσεως του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς. Αφορά κάποιον που όταν αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στη δημόσια διοίκηση, σαν δημόσιος υπάλληλο, προσλαμβάνεται με ένα μέτριο ποσό, αλλά ως διαμαγείας, μέσω αγνώστων διαδικασιών, στο τέλος της καριέρας, έχουν πολύ περισσότερα χρήματα. Ίσως σε κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κάποιοι να μην το γνωρίζουν αυτό στη νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου πέρασε αρκετό χρόνο, εργαζόμενος για την καταπολέμηση διαφθοράς, ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Δημόσιος υπάλληλος με πολύ μέτριο χαμηλό μισθό, ας πούμε 400 ευρώ το μήνα βγάζει, και όταν φεύγει μετά από μερικά χρόνια από την υπηρεσία του, έχει χιλιάδες ευρώ, να μην πω εκατομμύρια ευρώ και πολλά ακίνητα. Το 2003 η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κάλυψε το θέμα και προτάθηκε ότι τα συμβαλόμενα μέρη στη Σύμβαση εξετάζουν το ενδεχόμενο συμπερίληψη στο ποινικό δίκαιο νόμου διάταξης η οποία θα απαιτεί ένας δημόσιος υπάλληλος που δεν μπορεί να εξηγήσει το πόθεν έσχες της περιουσίας του ακριβώς να το εξηγήσει, να πει πόθεν έσχε. Όλα καλά και άγια. Υπάρχει προβληματάκι όμως. Κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπογράψει αυτή την ε, συγκεκριμένη διάταξη και πρόβλεψη. Και στην Ανατολική Ευρώπη μόνο μια χώρα το έχει συμπεριλάβει το μέτρο αυτό στην νομοθεσία. Το, η Μακεδονία, λέει ο μιλητή. με ενθάρρυνση ενό προγράμματο που υποστήριζε τη Βρετανία. Κρίμα διότι σε όλο τον κόσμο 44 χώρες, 44 χρησιμοποιούν αυτή την αρχή. Γιατί? Διότι μοιράζεται το βάρος. Το μοιράζεται το κράτος και ο κατηγορούμενος έχουν το βάρος απόδειξης. Για να αποδείξουν τα σοβαρότερα ποινικά δικήματα που γνωρίζουν αυτοί που ασχολούνται με το θέμα. Να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά με άλλα λόγια. Ποιο είναι το πρόβλημα με τη διαφθορά. Σπανίως υπάρχουν μάρτυρες. Θέλουν να, να πάνε στο δικαστήριο και να είναι μάρτυρες. Και το μόνο ίχνος που υπάρχει των δραστηριοτήτων, εκείνων που είναι παράνομοι, είναι η αύξηση, η ανεξήγητη αύξηση του πλούτου, της περιουσίας τους. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν αυτό το, αυτή την αρχή. Τη δεκαετία του 60 στη Λατινική Αμερική πρώτα εμφανίστηκε αυτή η αρχή και κυρίως στην Αργεντινή. Βέβαια μέχρι να εφαρμοστεί στην πράξη πέρασαν πολλά χρόνια. Το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποίησε αυτό το μέτρο τη δεκαετία του 70 και του 80 στο Χονγκ Κόνγκ. για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά του δημόσιου τομέα που μάστιζε το Χονγκ Κονγκ. Αποτελεσματικότατο μέτρο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως το αδίκημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρουν τι ισχύει. Καθένας είναι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίου, έχει δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, ε, διότι βασική είναι η αρχή που υπάρχει του καθήκοντος να εξηγεί κανείς πώς έχει δημιουργήσει την περιουσία του. Εγώ είμαι δημόσιο υπάλληλο και όλα τα μέλη της Επιτροπής που βλέπω μπροστά μου είναι δημόσιο υπάλληλοι. Πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία ενεργητικού, την περιουσία σας όταν αναλαμβάνετε τα καθήκοντα και να υπογράψετε τη δήλωση και να πείτε ότι είναι αληθής υπεύθυνη δήλωση είναι εν μέρη το καθήκον του να εξηγεί κανεί πώς δημιούργησε την περιουσία του. Εκτός, είναι διαφορετικό από ένα ποινικό αδίκημα απλό. Εάν η χώρα μπορεί να αποδείξει ότι ένα άτομο είναι δημόσιος υπάλληλο που ανέλαβε τα καθήκοντά του με ένα ποσοχή σαν περιουσιακό στοιχείο. Αυτό που αναφέρεται και στη δήλωσή του και αποχωρεί από την υπηρεσία με πολύ μεγαλύτερο ποσό, σαν περιουσία, εκείνοι πρέπει να αποδείξουν επαρκώς από πού προήλθαν τα χρήματα. Οι ορισμοί και οι έννοιες συζητούνται εκτενώς. Για τη σύντομη παρουσίασή μου όμως, μια ικανοποιητική εξήγηση εννοούμε κάποιον για τον οποίο είμαστε 51%. Ε, δηλαδή οι πιθανότητες είναι ότι αληθεύει η εικασία. Βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητείται κατά πόσο κάθε άτομο πρέπει να εξηγήσει οτιδήποτε. Έχω μόλις 11 λεπτά και δεν μπορώ να μακρηγορήσω κάποια μέλη της Επιτροπής των Επιτροπών, αν έχουν νομικό υπόβαθρο, θα, γνωρίζουν την έννοια αυτό να εξηγήσω την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Επιτρέπεται, σύμφωνα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν απαγορεύεται από κανένα σύνταγμα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Η υπόθεση αθωότητας δεν είναι κάτι απόλυτο, υπό όρους ισχύει. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι το αδίκημα, ο πυρήνας του αδικήματος χρησιμοποιείται αναλογικά, τότε καλύπτεται η υπόθεση της αθωότητος καθώς και η, πρόσβαση, η υπόθεση της πρόσβασης σε δίκαιη ε, δίκη. Μίλησα με την κυρία Ζολή για το θέμα αυτό. Στη Γαλλία ισχύει εξής αρχή. Μπορεί να αποδειχθεί ότι κάποιος που συνήθως έχει επαφές με οργανωμένους εγκληματίες και έχει τρόπο ζωής και χρήματα τα οποία δεν μπορεί να εξηγήσει, θεωρείται ότι είναι ένοχος ποινικού αδικήματος. Έπρεπε να μιλήσω γρήγορα, αλλά ελπίζω ότι μπορώ να βοηθήσουν οι διερμηνείς θα δείτε ότι υπάρχει μία ομοιότης, δηλαδή η απέτηση να δώσει εξηγήσει κανείς. Και για όλους μας, στο άλλο άκρο του φάσματος, αν αντιμετωπίσουμε έρευνα φορολογική, υπέχουμε καθήκον να εξηγήσουμε, αν γίνεται αυτή η έρευνα, το πόθεν έσχεσαι. έχουμε από τη μία πλευρά τη φορολόγηση που είναι πιο ριχά τα νερά και από την άλλη πλευρά τα πιο βαθιά νερά ποινική ε, νομοθεσία. Αυτές οι δύο επιτροπές εστιάζονται επί του εγκλήματος και της αναπτύξεως. Έθεσε το μόνο ερώτημα, κυρία Πρόεδρος. Τι γίνεται με τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Μερικά από αυτά πηγαίνουν στις τσέπες των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Να χρησιμοποιήσουμε έναν μηχανισμό όπως αυτόν που παρουσίασα. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίνινγκ. Πολύ περιεκτική και σύντομη παρουσίαση. Ο κύριος Μπέικερ έχει το λόγο να αναφερθεί στις ροές των παρανόμων πόρων. Είναι διευθυντής του Global Financial Integrity. Έχετε το λόγο. Ε, αν θέλετε πατήστε το κουμπί να ανοίξετε το μικρόφωνο. This one, Thank you. Thank you. Uh, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και έχω την ε, δυνατότητα να είμαι πάλι στην Επιτροπή της κυρίας ε, Ζολή. Το 1997 όταν ε, ταξίδευα να τον κόσμο και έπαιρνα συνεντεύξεις από διάφορους ανθρώπους όταν έγραφα το βιβλίο μου για τις παράνομες ροές ε, πήρα μια συνέντευξη από έναν Ελβετό τραπεζίτη στην Ελβετία και βεβαίως ε, του έδωσα την δικαίωμα τη ανωνυμία, έτσι ώστε να μιλήσει ειλικρινά και ανοιχτά μαζί μου και μου είπε ότι όσο τα χρήματα της ε, φοροαποφυγής δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τα χρήματα από τα ναρκωτικά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ξέπλυμα χρήματος και ακριβώς έθεσε το δάχτυλό του επί των τύπων των ύλων. Όσο κρατάμε ανοιχτό το σκιώδες οικονομικό σύστημα για να, να μην αντιμετωπίσουμε το θέμα της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι το σύστημα αυτό θα σταματήσει τις παράνομες ροές ή τις ε, ροές ε, χρημάτων από ε, διαφθορά. Είναι παγκόσμια η κίνηση των παράνομων αυτών ροών και βεβαίω επηρεάζουν πάρα πολύ τι αναπτυσσόμενες χώρες. Στην ανάλυση που κάναμε για το 2011 αναφέρονται 783 δισεκατομμύρια δολάρια που, που πηγαίνουν από τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες ε, παράνομα και χωρίς να καταγράφονται πουθενά. 783 δισεκατομμύρια λέει η ανάλυση μας. Ε, λίγο, λιγότερο, λίγο μικρότερο ποσό από τις αναλύσεις που είχαμε κάνει για τα δύο προηγούμενα χρόνια. Αλλά σκεφτείτε πώς έχουν φτάσει τα ποσά αυτά να είναι τόσο υψηλά ε, τα τελευταία χρόνια. Να έχουν φτάσει δηλαδή και σε, ε, σε, 3 εκατομμύρια, σε 3 που φεύγουν από τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Το Διεθνέ έγκλημα παράγει περίπου 650 δισεκατομμύρια δολάρια σε 12 κατηγορίες ε, παράνομων δραστηριοτήτων. Υπάρχουν και άλλε 12 κατηγορίες που δεν τι αναλύσαμε. Συμπεριλάβαμε όμως στην δική μας την ανάλυση και τα ναρκωτικά και τα, ε, την ε, παρανομή, το παράνομο εμπόριο ανθρώπων κτλ. Μιλάμε λοιπόν για εκατοντάδες εκατομμυρίων ή δισεκατομμυρίων δολαρίων τα οποία επηρεάζουν τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Πώς ρέουν τώρα αυτά τα κονδύλια περνάνε μέσα από σκιώδη οικονομικά συστήματα, τα οποία εμείς δημιουργήσαμε. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δεν είναι οι άνθρωποι στις χώρες αυτές από τις οποίες έρχονται τα χρήματα αυτά, που δημιούργησαν τα συστήματα αυτά, τα συστήματα τα ε, δημιούργησαν οι άνθρωποι από τις χώρες στις οποίες φτάνουν αυτά τα παράνομα ε, χρήματα. Και εδώ παίζουν ρόλο πολλά πράγματα, όπως ας πούμε φορολογική παράδειση. Όταν εγώ ξεκίνησα να εργάζομαι ε, στο, το, την δεκαετία του 60 υπήρχαν μόλις 4-5 ε, φορολογική παράδειση. Τώρα υπάρχουν περίπου 60 σε όλο τον κόσμο. Όλοι αυτοί οι φορολογικοί παράδειση λειτουργούν ως ε, μυστικές δικαιοδοσίες. Δηλαδή έχουν την υπονομή, έχουν τους τραπεζίτες, τους ε, λογιστές, τους οικονομολόγους, τους δικηγόρους που μπορούν να δημιουργήσουν κάποια κάποια, ε, κάποιες κατηγορίες πίσω από κάποια ψεύτικα ονόματα έτσι ώστε κανείς να μην ξέρει ποιος είναι τελικά ο κύριος ε, μέτοχος ή ο, ο κάτοχος αυτών των ε, ε, οργανισμών. Και βεβαίως μιλούμε για εκατομμύρια τέτοιους οργανισμούς ανά τον κόσμο. Επίσης, ε, ψεύτικες ψεύτικοι οργανισμοί ή πλαστά τιμολόγια χρησιμοποιούνται σε όλες τις ε, διαδικασίες ε, συναλλαγών, κυρίως στη χειραγώγηση τιμών, στις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι περίπου 60-70% των παράνομων χρημάτων που περνούν τα σύνορα προκύπτουν από εμπορικές δραστηριότητες. Το έγκλημα που είναι και αυτό βεβαίως ένα κομμάτι του θέματος που συζητούμε σήμερα, οι, οι ε, εγκληματικέ δραστηριότητε ε, κατέχουν μόνο ένα 30-35% του μεριδίου αυτών των διασυνοριακών ε, μετακινήσεων. Τα λεφτά που κλέβονται, που μέσω ας πούμε κλοπής υδροδοκίας των διοικητικών υπαλλήλων φτάνουν μόλις το 5% του παγκοσμίου συνόλου. Ένα ακόμη στοιχείο του συστήματος αυτού που μεταφέρει χρήματα ανά τον κόσμο είναι διάφορες τεχνικές ξεπλήματος που χρησιμοποιούνται κυρίως για ειδικού σκοπούς. Και βεβαίως υπάρχουν και πολλές, πολλοί νόμοι που βεβαίως διευκολύνουν την διακίνηση αυτών των χρημάτων μέσω των σχεδόν αυτών οικονομικών συστημάτων και τα οδηγούν στις δυτικές οικονομίες. Υπάρχουν λοιπόν κενά και στις δικές μας ε, νομοθετικές ρυθμίσεις. Έχουμε βλακεί ε, στην, ε, πολύ σημαντικά στην αντιμετώπιση του ξεπλήματος, μαύρου χρήματος, από ναρκωτικά, από έγκλημα εδώ και 20 χρόνια. Δεν τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε αποτύχει. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι η αύξηση του, του ε, μαύρου χρήματος αρχίζει, είναι ότι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μάλλον αρχίζει να μειώνεται. Το κάθε άλλο παρά. Φαίνεται ότι συνεχίζει να αυξάνεται. Τα ναρκωτικά δεν έχουν μειωθεί, ούτε σε όγκο, ούτε σε τιμή, ούτε σε αξία. Το διασυνοριακό έγκλημα άλλου είδου επίσης έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία 20 με 25 χρόνια το, η βασική αποτυχία σε, αυτό το, σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε παγκοσμίω για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος είναι ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τη χρήση αυτών των σκιωδών οικονομικών συστημάτων για να μετακινήσουμε τα χρήματα της φοροδιαφυγής κάνοντας όμως κάποιους να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα δικά του συστήματα για να μετακινούν χρήματα από διαφορά ή από εγκληματικέ δραστηριότητε. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό είναι ένα θέμα όπου μπορούμε να επιτύχουμε μόνο εάν όλοι αναλάβουν την ευθύνη τους στο πρόβλημα. Έχει λοιπόν αλλάξει το κέντρο βάρους τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον για εσά εδώ στην Ευρώπη, παλαιότερα οι ΙΠΑ είχαν αναλάβει τον ηγετικό ρόλο για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Ε, πέρασαμε και μια νομοθεσία σχετική το 1977 που ήταν παράνομο να, που ήταν παράνομο δωροδοκεί κανεί ξένου ε, δημοσίου υπαλλήλους. Ξεκινήσαμε κάποιες νομοθεσίε ε, το, τη δεκαετία του 80 για την αντιμετώπιση του ξεπλήματο. Ενθαρρύναμε τη δημιουργία του G, μάλλον G7 να δημιουργήσει ε, ένα παγκόσμιο φορέα παρά, ε, αντιμετώπισης της, ε, του ξεπλήματος μαύρου χρήματος που έγινε μια σχετική task force αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα έχει αναλάβει τα ενία για αυτά τα πράγματα και βεβαίως έχουν γίνει πάρα πολλά θετικά βήματα μέσω οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέσω άλλων δραστηριοτήτων που έχετε αναλάβει εσείς. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο τομείς όπου νομίζω ότι μπορούμε να προοδεύσουμε ακόμη περισσότερα όπου μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Αυτές, αυτοί οι δύο τομείς είναι η ιδιοκτησία και η, η φοροδιαφυγή. Καταρχάς, ποιοι είναι αυτοί που κατέχουν λογαριασμούς. Πρέπει να βρούμε. Να ξεκινήσω για αυτό λέγοντας ότι δεν υπάρχει ε, κανένα επιχείρημα υπέρ του να μην ξέρει κανείς με ποιον συναλλάσσεται. Δεν υπάρχει επιχειρηματολογία υπέρ του να μην γνωρίζεις. Δεν ποια είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τους λογαριασμούς με τους οποίους ασχολούμαστε. Και βεβαίως υπάρχουν εκατομμύρια επί εκατομμυρίων λογαριασμοί σε δικά σας σε τραπεζικά ιδρύματα, στα δικά μας, για τα οποία δεν ξέρουμε ποια είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αυτούς τους λογαριασμούς. Ε, ε, στα, στο υλικό που έχω ε, μελετήσει δεν βλέπω κανέναν τρόπο αποτροπής δημιουργίας κάποιων άλλων ανώνυμων εταιριών ή ανώνυμων λογαριασμών. Και θα ήθελα να προτείνω δύο τρόπους με τους, με τους οποίους θα μπορούσαμε ίσως να παρέμβουμε νομοθετικά για να ε, λύσουμε το πρόβλημα. Καταρχάς, για αυτές τις ε, ιονί εταιρείε. Ας τις ε, κηρύξουμε παράνομες. Είναι ακραίο αυτό. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, το Κογκρέσο πέρασε το, την, το Patriot Act στο οποίο περιλαμβάνεται ένας, μια πολύ σημαντική ενισχυμένη, ένα σημαντικό κομμάτι ενισχυμένο για την αντιμετώπιση της της φοροδιαφυγής με Ιωνίοι τραπεζικές, τραπεζικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούσαν ε, ε, με ψεύτικα στοιχεία χωρίς να ξέρει κανείς ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις τράπεζες. Και το Patriot Act λέει ότι είναι παράνομο για οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό αμερικανικό ίδρυμα να λάβει χρήματα από ξένη τέτοια τράπεζα. Επίσης λέει ότι είναι παράνομο για οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του κόσμου να στείλει χρήματα στην, στις ΗΠΑ που έχει λάβει το ίδιο από κάποια άλλη ιονή τράπεζα ε, έτσι ώστε να αποφύγουμε να υπάρξει μεταφορά χρημάτων από, από κάποια χώρα προς τη Νέα Υόρκη πριν αυτά τα χρήματα φύγουν από τη Νέα Υόρκη και πάνε αλλού. Ε, όταν λοιπόν πέρασε το Patriot Act στη ΣΥΠΑ, αυτά τα ιδρύματα έκλεισαν σε όλο τον κόσμο. Από χιλιάδε που υπήρχαν, έφτασαν να μετρώνται στη ε, δάχτυλα του ενό χεριού εν μία νυχτή. Ήταν θέμα πολιτική βούληση των ΗΠΑ για να λύσουν αυτό ακριβώ το πρόγραμμα του σκιώδους οικονομικού συστήματος. Ακόμη υπάρχουν βεβαίως ελάχιστες τέτοιες τράπεζες που, που λειτουργούν στην Ευρώπη και θα πρέπει να ελέγξετε τις ε, δραστηριότητες τους έτσι ώστε να μην φτάσει κανένας, καμία από τις δραστηριότητες τους σε ε, λογαριασμούς στις ΕΠΑ. Αλλά σχεδόν εξαφανίσαμε αυτές, αυτές του είδους τις ε, τράπεζες. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τις ιονί εταιρείε. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αν τώρα αυτό είναι πολύ ακραίο, υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος για την εξέβρεση των ιδιοκτητών των λογαριασμών. Είναι τα ε, δημόσια μητρώα για το ποια, ποιοι είναι οι κάτοχοι, ποιοι είναι οι πρόεδροι των επιχειρήσεων, ποιοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αυτούς τους λογαριασμούς. Αυτά μπορούν να καταγράφονται σε δημόσια μητρώα οι εταιρείε δημιουργούνται από κάποιε. Ε, από, μάλλον το κράτο έχει δικαίωμα να ξέρει ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτέ τι εταιρείε και βεβαίω οι πολίτε του οποίου εκπροσωπεί το κράτο έχουν το δικαίωμα να ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που κατέχουν αυτέ τι ε, ε, εταιρείε. Αυτά λοιπόν τα δημόσια μητρώα είναι άλλο ένας τρόπος να καταγράφονται οι κάτοχοι των λογαριασμών αυτών. Μετά, το επόμενο σημείο για το οποίο θέλω να σας μιλήσω ήταν, είναι η ε, φοροδιαφυγή, η φοροαπάτη. Το μεγαλύτερο κομμάτι της φοροαπάτης έχει να κάνει με ε, ε, τιμολόγηση και λαθασμένη τιμολόγηση εμπορικών συναλλαγών μεταξύ διαφόρων μερών που γίνεται για να αλλάζουν οι, εισαγωγές, ε, οι τιμές εισαγωγών και εξαγωγών στις συμπορικές δραστηριότητες για να μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί τον, τους ειδικού φόρους κατανάλωσης, το ΦΠΑ ή άλλα είδη εσόδων που θα έφταναν κανονικά στα κρατικά ταμεία. Στη ΣΥΠΑ αποφασίστηκε από το Ανώτερο Δικαστήριο το 2005 για μια υπόθεση ε, ε, είπα απέναντι στους, στον Πασκουαντίνο ο οποίος ήθελε να φέρει ε, παράνομο ε, αλκοόλ από τη ΣΥΠΑ στον Καναδά. Το ανώτερο δικαστήριο αποφάσισε ότι αυτό ήταν κόλπο για να υπάρξει απάτη. Το ενδιαφέρον με αυτή την υπόθεση Πασκοντίνο ήταν ότι δεν βασίστηκε στο ποιος τελικά ήταν αυτός που έχασε, που ουσιαστικά ήταν η καναδική κυβέρνηση, ή τι ακριβώς ε, χάθηκε, ήταν τα, οι τελωνιακοί δεσμοί. αλλά είπαν ότι έχετε ε, εγκατασταθεί στις ΕΠΑ και έχετε εμπλακεί σε ένα σχέδιο για να εξαπατήσετε. Και αυτό ε, αποφάσισε, η, αυτό, έτσι αποφάσισε, έτσι έκρινε το ανώτερο δικαστήριο. Σκεφτείτε πόσες αποφάσεις του ίδιου διαμετρήματος λαμβάνονται κάθε, κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο. Αποφάσεις ε, για την ε, ε, αντιμετώπιση της φοροαπάτης, της κατάχρησης του ΦΠΑ, της, των ειδικών φορών κατανάλωσης, είτε στην χώρα εισαγωγής, είτε στην χώρα εξαγωγής σε εμπορικές συναλλαγές. Όταν οι διοικητέ των εταιριών ξεκινούν τέτοιες δραστηριότητε, κάνουν ποινικό δίκημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, στις, ε, να το ξεκαθαρίσετε εσείς στις προτάσεις νομοθεσίας σας. Η απάτη θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Σημαίνει ε, παράνομη τιμολόγηση και λανθασμένη τιμολόγηση εμπορικών ε, εμπορευμάτων μεταξύ αρχών, έχοντας ως στόχο να καταχραστεί κανείς τα, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των ε, ΦΠΑ και, άλλες, ε, και άλλα χρήματα. Θα σας ενθάρρυνα λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, σκεφτεί την ενίσχυση αυτών των δύο πτυχών στην νομοθεσία που έχετε. Τους ιδιοκτήτες των λογαριασμών και το θέμα της φοροαπάτης. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Μπέικερ για την παρουσίασή σας. Πολύ σημαντικά τα επιχειρήματά σας. Στην ε, Επιτροπή ΚΡΙΜ θεωρήσαμε και εμείς ότι δεν πρέπει να διαχωριστούν τα χρήματα που ε, προκύπτουν από, την, ε, από το έγκλημα, από τα χρήματα που προκύπτουν από την φοροαποφυγή που γίνονται μέσω διαφόρων εταιριών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλάζω μικρόφωνο, συγγνώμη. Πάμε τώρα στην κυρία Jennifer Bramlett. από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα του ΙΕ για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης ε, του, της τρομοκρατίας. Έχετε και εσείς 15 λεπτά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και να προλαλήσατε για τα εξαιρετικά πράγματα που μας είπε. Ίσως ε, επαναλάβω κάποια από αυτά που είπε, αλλά θα ζητήσω την υπομονή σας γιατί όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Μια ε, γνωστή ρίση λέει ότι το έγκλημα αποδίδει. Και υπάρχει μια αλήθεια γιατί αν δεν μπορούσαν να κερδίσουν οι εγκληματίε δεν θα έκαναν εγκληματικέ ενέργειε. Και ο τρόπο προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι θα εξακολουθεί να αποδίδει το έγκλημά του ε, οι εγκληματίε είναι ακριβώ το ξέπλυμα χρήματο. Γιατί καλύπτοντα την προέλευση ε, των εσόδων του μπορούν να αποφύγουν την, την οντοπισμό και την περίπτωση να διωχθούν αν μετά τα δαπανίσουν ή τα επενδύσουν κάπου. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ρίση ότι δεν αποδίδει το έγκλημα και αυτό ε, μπορούμε να το περάσουμε ως μήνυμα αν επιτεθούμε στις ροές από τους ε, εγκληματίες. Μπορούν να αποσταθεροποιήσουν τα κράτη αυτούς που ε, καταφεύγουν στις εγκληματικές δραστηριότητες επηρεάζοντας και τον, την, την προσέλκυση νέων και μειώνοντας το κέρδη τους. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε λοιπόν ε, τις παρανόμες ροές μεταξύ αυτών ε, χρωματοδότης τρομοκρατίας, ε, ξέπλυμα χρήματος κτλ. Πολλά στρώματα υπάρχουν. Το σημαντικότερο βήμα που πρέπει να κάνει μια χώρα, που μπορεί να κάνει, είναι να έχει ένα καθεστώς καταπολέμησης της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με νόμους, κανονισμούς που συμμορφώνονται με τα διεθνή αποδεκτά πρότυπα. Έχουμε πολλά τέτοια, όπως είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, η Σύμβαση κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος και έχουμε και τις 40 ε, συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης, ε, FAT FIGAF, όπως είναι γνωστή. Θα πρέπει όμως κυρίως να υπάρξουν σαφές ποινές για αυτό το έγκλημα της ξεπλήματος χρήματος. Θα πρέπει να υπάρχουν διατάξεις για το πάγωμα και την κατάσχεση των ε, περιουσιακών στοιχείων που έρχονται από και δραστηριότητα. Θα πρέπει να ε, υπάρξει νομοθεσία λοιπόν στις χώρες για να μπορούν και να ανακτούν τα δημευθέντα αυτά κονδύλια. Πρέπει λοιπόν η νομοθεσία να περιλαμβάνει και διατάξεις για τη διεθνή συνεργασία, αμοιβαία δικαστική συνδρομή, έκδοση και άλλες μορφές δικαστικής συνεργασίας. Επίσης, απαιτούνται διάφορες πρακτικές, ιδέουσα, ιδέουσα επιμέλεια, η καταγραφή κτλ. Και μια άλλη ε, σημαντική υποχρέωση είναι αυτή της, του reporting, της καταγραφής. Δηλαδή, ε, οι μεσίτες, οι έμποροι ε, πολύτιμων ειδών, οι, παραδείγματος χάρη χρυσού, ή διαμαντιών, θα πρέπει να συνεργάζονται με τις αρχές, να δίνουν όλες τις πληροφορίες. Θα πρέπει να υπάρχει επίση και μια στεναρή φορολογική πολιτική. Αποτελεσματική έλλειψη στα σύνορα είναι απαραίτητη επίση για να μην υπάρχει λαθρεμπόριο υψηλών, υψηλής αξίας αγαθών ή χρημάτων. Επίσης, οι ανεπίσημοι οργανισμοί ή τα ε, αγαθοεργή ιδρύματα θα πρέπει να ελέγχονται στις συναλλαγές. ένα επόμενο βήμα για τον έλεγχο και τον περισμό των παράνομων οικονομικών ε, Ρόν είναι πώς θα λειτουργεί, ε, με τι προτεραιότητες θα λειτουργεί. Έχουμε την ε, μονάδα οικονομικών πληροφοριών και πολλές άλλες αρχές που θα πρέπει να συνεργάζονται για να δείχνουν περιπτώσεις ε, χρηματοδότησης τρομοκρατίας, ξεπλήματος χρήματος, να παρακολουθούν τα ίχνη του χρήματος αυτούς για να μπορούν να εντοπίζονται, να ερευνώνται, να παγώνουν και να κατάσχονται ε, τελικά αυτά τα χρήματα και να μπορούν ενδεχομένως μετά και να τιμωρηθούν αφού βρεθούν οι ένοχοι. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχουν και οι κατάλληλοι θεσμοί ποινική δικαιοσύνη και ότι ε, έχουν και την εξουσιοδότηση για να εφαρμόσουν του κανονισμού για το ξέπλωμα ε, βρώμικου χρήματο. Έχουν το απαραίτητο προσωπικό με τι δεξιότητε και τη στήριξη την απαραίτητη για να φέρουν σε πέρα τη δουλειά του. Επομένω, η δημιουργία υποδομών και η εκπαίδευση είναι κάτι πολύ σημαντικό ε, και σίγουρα η πολιτική βούληση διαδραματίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλους αυτούς τους τομείς. Είναι πάρα πολύ απαραίτητο και η αστυνομία να έχει ειδική ε, εκπαίδευση για το πώς θα διεξάγει αυτές τις οικονομικές έρευνες, γιατί χρειάζονται διαφορετικές δεξιότητες για αυτή την, του είδους την έρευνα, πρόσβαση, κατανόηση ε, ειδικών πληροφοριών είναι κάτι διαφορετικό από τη διαρρεύνηση μια κλοπή ή ενός φόνου. Επίση θα πρέπει να υπάρχει δραστηριότητα μεταξύ εισαγγελέων, ανακριτών, ε, τη υπηρεσία οικονομικών πλοίων κτλ. Γιατί με αυτή τη συνεργασία οι ερευνητέ ε, θα μπορούν να δημιουργήσουν και κάποιες αλυσίδες αποδείξεων στοιχείων για να μπορέσουν να οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη δίωξη των εγκληματιών. Πρέπει να υπάρχει επίσης και ε, σε εθνικό επίπεδο συνεργασία εμείς καλούμε πολλές φορές και επαγγελματίε από διάφορους κλάδους σε επιμορφωτικά σεμινάρια για να υπάρχει ε, μία επιμηξία και αλληλό μετάδοση γνώσεων. Και ο ιδιωτικό τομέα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει, όπω και αυτοί που έχουν ε, τι ε, αρμοδιότητε στον τομέα του reporting, να παίρνουν και αυτοί αυτή την εκπαίδευση. Δεν θα πρέπει επίσης ε, να ξεχνάμε ότι και η καλή περιφερειακή συνεργασία είναι αποτελεσματική στην καταπολέμηση ε, αυτών των εγκλημάτων, γιατί οι εγκληματίες δεν γνωρίζουν σύνορα και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα να συνεργάζονται μέσω συνδικάτων παγκοσμίων. Και έτσι και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται πέραν των σύνορων, να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και να κάνουν κοινέ επιχειρήσεις. Ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις έρευνες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματο είναι το κύριο έγκλημα, πρέντι και το φένς. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δικήματα, κάποιε αξιόπινε πράξει από τι οποίε ε, μετά ξεπλένεται χρήματα από απάτη, διαφθορά. Αλλά ε, σε λίγε χώρε περιλαμβάνεται στον ποινικό κώδημα ω από μόνο του έγκλημα, ω από μόνο τη αξιόπινη πράξη, το ξέπλυμα του ε, βρώμικου χρήματο. Και θα πρέπει να εξετάζεται το κύριο έγκλημα που δεν είναι στην περίπτωση αυτή το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Θα πρέπει να γίνει μια μετατόπιση, μεγάλη μετατόπιση και εμείς πιστεύουμε ότι οι αρχές θα πρέπει άμεσα να ξεκινούν παράλληλες ταυτόχρονες έρευνες ε, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές ροές ε, προσόδων από κλιματικές δραστηριότητες να ξεκινούν έρευνα για κάποιο κύριο έγκλημα. Το να παρακολουθεί κανείς τα χρήματα μπορεί ε, να βρει περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα έπρεπε και θα μπορούσαν να δημευθούν και οι εγκληματίες που συμμετέχουν θα μπορούσαν να δικαιωθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Όλα αυτά είναι λογικά και ωραία στα συστήματα που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες αλλά μου ζητήσατε να μιλήσω για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος ε, και του ξεπλήματο χρήματο στι ανεψόμενες χώρες. Πρέπει να σας πω ότι ναι, ουσιαστικά είναι οι ίδιες οι βασικές δομές, θα πρέπει να ε, προσαρμοστεί η εφαρμογή του είναι ηλεκτρονικά τα χρηματοοικονομικά συστήματα σε μεγάλο βαθμό, οπότε εμείς έχουμε πολλές μορφές ε, ταυτοποίησης, αναγνώρισης. Έχουμε ε, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, συστήματα τεχνολογίας των πληροφοριών και μηχανισμούς που μπορούν να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών όπως επίσης και την περιφερική και διεθνή συνεργασία. Έχουμε χιλιάδες εκπαιδευμένο προσωπικό. Παρά τα αυτά όμως ε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια χώρα η οποία ε, θεωρείται ότι συμμορφώνεται πλήρως σε όλες τις κατηγορίες που μελετά η ΦΑΤΦ αυτή η δική ομάδα ε, και ε, υπάρχουν μειονεκτήματα. Τι προκλήσεις λοιπόν αντιμετωπίζουν οι ανεψόμενες χώρες ό,τι αφορά τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Θα σας αναφέρω κάποια θέματα τα οποία τα εντοπίσαμε στις, ε, στα διάφορα εργαστήρια που είχαμε σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και κάποια από αυτά μας τα έχουν επισημάνει οι ίδιες οι χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζει ο πληθυσμός τον κίνδυνο των ε, χρηματοοικονομικών όρων, των παράνομων. Πολλές φορές έχουμε μεγάλα χρήματα τα οποία ε, μεταφέρονται με εμβάσματα και αυτό θεωρείται πάρα πολύ λογικό. Πολλές ανεψόμενες χώρες έχουν ε, οικονομίες που βασίζονται στα μετρητά. Και πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Άρα μετακινούν ε, από μόνοι τους τα χρήματα, τα μετρητά. Ή χρησιμοποιούν ε, άτυπες μορφές, τα χαβάλα ή άλλα συστήματα που δεν μπορούν να εμπέσουν στο, στη ρυθμιστική δυνατότητα τη τηλεφωνική, στις τηλεφωνικές ή ε, ε, ε, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές μέσω του κινητού ή του τηλεφώνου μπορεί κανείς χωρίς μεγάλο κόστος να κάνει τραπεζικές συναλλαγές. Αυτές οι συναλλαγές δεν μπαίνουν όμως στις απαιτήσει του να γνωρίσει κανείς τον πελάτη και στη δέωση επιμέλεια και δεν αναζητούνται ε, οι ύποπτες συναλλαγές. Επίσης δεν υπάρχουν σε πολλές χώρες συστήματα για την έκδοση ε, ταυτοτήτων. Και σε πολλές χώρες ε, θεμητά νόμιμα μπορεί κανείς να έχει πολλά ονόματα. Άρα δύσκολο είναι να ξέρει κανείς ποιος ανοίγει ένα οργανισμό ή ποιος ε, μεταφέρει κάποια χρήματα. Υπάρχουν πολύπλοκα συστήματα δεδομένων. Ε, αυτά όμως είναι ε, δύσκολα γιατί δεν επιτρέπουν την καταγραφή και την διατήρηση αρχείων από τους αξιωματούχους. Σε πολλές ανθρώμενες χώρες οι ειδικοί δεν έχουν επίσης πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο ή σε λογισμικό AML ούτε την ικανότητα να αναζητήσουν νέες μεθόδους εμβασμάτων μεταφοράς χρημάτων. Πολλοί έχουν κάποιους τρόπους ε, μεν ε, επικοινωνίας, αλλά όχι αξιόπιστες μεταξύ των διαφόρων φορών. Ούτε και αξιόπιστη νομοθεσία AML έχουν πολλές χώρες. Ούτε και την πολιτική βούληση να τη δημιουργήσουν και να την εφαρμόσουν. Υπάρχουν 15 ε, δικαιοδοσίες στις δημόσιες δηλώσεις ε, της FATF, blacklist, μαύρη λίστα όπως λέγεται. Και υπάρχουν και στην κρίζα και αρκετά σκούρα λίστα ε, άλλες πολλές χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ε, δημιουργεί εμπόδια στην καταπολέμηση των παράνομων και μπορούν οι χώρες με διάφορους τρόπους να βελτιώσουν την προσπάθειά τους. Έχουμε ένα πρόγραμμα κατά της χρηματοδότησης της GPML λέγεται, και εδώ και 15 χρόνια βοηθάμε στην καταπολέμηση του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο. Είχαμε επιτυχίε σε πολλούς τομείς. Ανέφερα ε, την επιμόρφωση εξωματούχων με ε, δραστηριότητα στον τομέα του reporting ε, κτλ. ή στον τραπεζικό τομέα. Πάντω σε αναψώμενες χώρε υπάρχουν κάποιε κυβερνήσεις που έχουν δημιουργήσει πολιτικέ όπου παραδείγματος χάρη οι αξιωματούχοι παίρνουν το μισθό τους ε, σε ένα τραπεζικό λογαριασμό ή μειώνονται ε, τα οι επιβαρύνσεις για να προσεγγιστούν περισσότεροι πελάτες και για τη Χαβάλα γίνονται προσπάθειες να εφαρμόζει κάποια πρότυπα. ενημερώνονται αυτοί της Χαβάλα αλλά και άλλων άτυπων δικτύων μεταφοράς χρημάτων για τις υποχρεώσεις που έχουν να τηρούν παραδείγματο χάρη κάποια αρχεία και ούτω καθεξής. Εμείς στη Σομαλία και στην Αιθιοπία σύντομα θα προβούμε σε ε, επιμόρφωση και επίσης ε, θέλουμε οι κυβερνήσεις ε, να προβαίνουν και σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η δραστηριότητα ξεπλήματος χρήματος, το οικονομικές ροές. Και έχουμε ειδικά προγράμματα για τις συνθήκες της κάθε χώρας. Από τα πιο απλά στα πιο προηγμένα. Όταν δηλαδή ε, δεν υπάρχουν ε, προγράμματα λογισμικά μπορεί να βοηθήσει με την οικονομική ε, ομάδα Δεν υπάρχουν όμως μόνο τεχνικές ε, δεξιότητες που είναι απαραίτητες και τη δομική σκέψη, την κριτική σκέψη, την επίλυση ε, προβλημάτων προωθούμε με προγράμματά μας. Έχουμε επίσης ε, και κάποιους εμπειρογνώμονες στον τομέα AML σε πέντε περιοχές του κόσμου που βοηθούν καθημερινά. Σε πολιτικό επίπεδο ενθαρρύνουμε τις χώρες να τηρούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών συνθήκων και να παρέχουν το πλαίσιο για την αναζήτηση κοινών λύσεων. Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα νωρίτερα στην ε, παρουσίασή μου, που είναι και τα θεμέλια για την ε, καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και του, διεθνούς, του οργανωμένου εγκλήματος σε όλες τις δικαιοδοσίε των αναπτυγμένες όχι. Δηλαδή, δημιουργία καθεστώτων για την αντιμετώπιση της, ε, του ξεπλήματος βρώμικου χρηματιστώσεων δημιουργία των υποδομών για την ανάλυση, τον εντοπισμό, τη δίμευση των παράνομων περιουσιακών στοιχείων. Με όλα αυτά και με άλλα μπορούν τα κράτη να ανακτήσουν τον έλεγχο και να αποσπάσουν από τις εγκληματίες ε, τις παράνομες προσόδους τους, γιατί έτσι τους χτυπάμε εκεί που πονούν περισσότερο, στην τσέπη τους, στο πορτοφόλι τους. Σας ευχαριστώ και είμαι στη θέση σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Thank you very much. Ε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Έχουμε τον κύριο Γιακολίνο τη Ειδική Επιτροπή, τον εισηγητή των Προσύνων, και έχουμε και τον εισηγητή πόλη τρομοκρατία και ε, κατά πολέμηση ξεπλήματο χρήματο, την κυρία Σαζωτίνη και τον κύριο Γκόμε, που ετοιμάζει έκθεση διαφθορά. Δίπλα μου εδώ στην Προεδρία είναι η συντάκτρια τη ε, ε, γνωμοδοτήσεω ΔΕΒΕ για την έκθεση ΚΡΙΜ και συζητούμε τώρα για την διάμεση έκθεση τη ειδική Αρμόδης Επιτροπή. Άρα κάθε πρόταση είναι πρόσδεκτη. Πριν δώσουμε το λόγο, στους ευρωβουλευτές. Ίσως θα ήταν καλό να ακούσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί της καταστάσεως νέες προτάσεις στον τομέα αυτό. Κάποιος από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα ήταν σε θέση να πάρει το λόγο. Ο κύριος Γέσπι Πέντερσον από την ΤΕΦΚΟ μπορεί να πάρει στο λόγο να μας πει μερικά πράγματα. Τι ακριβώς γίνεται στον Περλιμού. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι, λέγομαι Βαντεμίρ. Είμαι το πρόγραμμα για το εργαλείο για την σταθεροποίηση. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη σημερινή συνεδρίαση η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε κάποια κίνητρα για να γίνει η δουλειά πρέπει να γίνει. Όσον αφορά αυτό το μέσο για τη σταθερότητα, στα πλαίσια αυτού έχουμε δρομολογήσει προγράμματα στον τομέα της καταπολεμήσεως του οργανωμένου εγκλήματος και σχετικά με αυτό εστιάζουμε τις δραστηριότητές μας βασικά στην καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, καταπολέμηση λαθρεμπορίου ανθρώπων και ούτω καθεξής. Οπότε δεν έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα με στόχο την καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, χρήματος, εστιαζόμεθα επί προσπαθειών αποθάρρυνσης του εμπορίου στους τομείς που προανέφερα. Άρα ε, καταπολεμούμε την κοκαίνη και την ερωίνη και τις διαφρομές μεταφοράς τους Άλλαξε η κατεύθυνση, οι διαδρομέ που ακολουθούνται, γίνεται όλο και πιο σημαντική η διαδρομή μέσω Αφρικής. Διότι δεν υπάρχει επαρκής οικονομικός έλεγχος εκεί, πιστεύουμε. Και τέλος, εξίσου σημαντικό, άλλα συνθετικά ναρκωτικά, άλλα προϊόντα διακινούνται τώρα. Εξετάζοντας λοιπόν το παράνομο εμπόριο παρανόμων προϊόντων, σαν παραπροϊόν εξετάζουμε και το πώς θα ενισχύσουμε τα διάφορα συστήματα καταπολεμήσεως της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων στα διάφορα κράτη, τούτων λεχθέντων. Όταν θα εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2014, θα προσπαθήσουμε να δρομολογήσουμε κάποια προγράμματα κυρίως στις αφρικανικές χώρες, ούτως ώστε να ενισχύσουμε τα συστήματά τους. Αυτά που έχουν διαπιστώσει και αρμόδιοι φορείς του ΟΗΕ για να θεσπιστεί κατάλληλη νομοθεσία και να δημιουργηθεί και το κατάλληλο διοικητικό δυναμικό, να επιβληθεί ο νόμος και να αυξηθεί περαιτέρω δυνατότητα κατάσχεσης παρανόμων προϊόντων και να, να καλύψουμε τις διάφορες πτυχές. Εδώ βρισκόμαστε, πρώιμο στάδιο. Υπάρχουν πολλές άλλες προτεραιότητες. Όσον αφορά τις χώρες γειτονίας, προσπαθούμε να εθετήσουν οι χώρες το κεκτημένο το κοινοτικό και να γίνουν εναγκαίες διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Εν γέννη, ειλικρινά, ανάμεικτη εικόνα. Οπότε καλωσορίζουμε εκδηλώσεις όπως η παρούσα για να μας βοηθήσουν να καθορίσουμε εξωτερικά προτεραιότητες. Ευχαριστώ κύριε Βαντεμίρ. Αρκετοί έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ τους συναδέλφους να αυτοπεριοριστούν σε δύο το πολύ τρία λεπτά για κάθε παρέμβαση. Ο κ. Γιακολίνο, ε, που είναι συγητής της Ειδική Επιτροπής ΚΡΙΜ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Πρόεδρο Ζολή. Ακούσαμε με τα ζωηρού ενδιαφέροντος τις ε, παρεμβάσεις από τους δύο συγητές. Το θέμα του ξεπλήματος χρήματος είναι ένας τομέας που αφαιρεί πολλούς πόρους από την νόμιμη οικονομία. Υπάρχει δίσδυση των εγκληματικών οργανώσεων που εκμεταλλεύεται τα χρήματα. Ξεκινήσαμε μια δουλειά που έχει φτάσει σε καλό σημείο. Χθε παρουσιάστηκε η έκθεση ενδιάμεση. Όταν η κυρία Μπέικερ είπε ότι υπάρχουν ακόμα 60 φορολογικοί ε, παράδεισοι, είπε ο κ. Μπέικερ μάλλον, ε, δείχνει πόσο αναγκαία είναι συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Και υπάρχουν 783 δισεκατομμύρια που περνούν από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σκέψεις και ερωτήσεις. Προς τον κύριο Μπέικερ Ελπίζω να μας ακούει, να μ' ακούει και ο Μπέικερ. Ο οργανισμός σας εδρεύει στην Ουάσιγκτον, κύριε Μπέικερ. Απ' την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, του κόσμου θα έλεγα. Στην άλλη άκρη του κόσμου έλεγε και ο Πάπας ε, Φρανσίσκος. Έχουμε όμως πολύ στενές εμπορικές σχέσεις ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείες και έχουμε συνάψει και συμφωνία. Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Πόσο μπορεί να χρησιμεύσει για την καταπολέμηση του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο και η ανάλογη συμφωνία με τον Καναδά. Αυτέ οι οικονομικέ ροέ μπορούν να ελεγχθούν επαρκώ μέσω των εμπορικών συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ΗΠΑ, παραδείγματο χάρη θα μπορούσε να είναι σημαντικότατη πειραματική συμφωνία. Προς τη κυρία Μπράμλετ μας λέει και σωστά ότι πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία. Και στι αναπτυσσόμενε χώρες ποτέ δεν, μάλλον δεν υπάρχει σωστή αντίληψη όσον αφορά την παρανομή ροή χρημάτων. Χρειάζονται προληπτικοί έλεγχοι. Χρειάζεται έλεγχος, προσμέτρηση, ερώτηση. Υπήρξαν περιπτώσεις ξεπλήματος που ανακαλύψατε σε ποιες χώρες, μπορούμε να το ξέρουμε. Ποιος ο ρόλος των ΜΚΟ που ίσως και εν αγνία τους ενεπλάκησαν κατά κάποιο τρόπο σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι υπερεθνικό αδίκημα το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και για να αντιμετωπιστεί επαρκώς χρειάζεται μεγάλη νομική συνεργασία, αστυνομική συνεργασία και ίσως να βοηθούν και διάφορες συμφωνίες με τρίτες ε, χώρες. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Μίτσελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τον αναπτυσσόμενο χώρο, τι προσδοκίες υπάρχουν όταν αυτοί βλέπουν τι γίνεται στον αναπτυγμένο κόσμο. Πολύ μεγάλο ερώτημα, αλλά θα πρέπει να ξαναμπεί ο όρος κοινωνικός στην, κοινωνία, στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει χειραγώγηση, αναλαμβάνεται ο κίνδυνος από διοντολογικά σωστά, να μην υπάρχει ε, έλεγχος Καμιά φορά, αν δεν, υπάρχουν, αν δεν, δεν, αν δεν υπάρχει σωστή ιδεοντολογία όσον αφορά τη λειτουργία τη αγορά, είναι θέμα ηθικό αυτό. Πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Καλύτερα να βγάζουμε χρήματα από τα ναρκωτικά παρά από κάποιε θεμητέ, όπω αποκαλούνται εμπορικέ πρακτικέ. Έχουμε στην Ιρλανδία αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση των στοιχείων ενεργητικού για πορέπτο έγκλημα. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει ποινικό μητρό ή όχι. Γίνεται με βάση το αστικό δίκαιο. Αν υποθέτει ο νόμο ότι έχει κάποια χρήματα που δεν πάει τα δικαιολογήσει, μπορεί να τα κατάσχουν και εσύ πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι παράνομο. Και αυτό το εξετάζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά το Κοινοβούλιο, έχουμε προσπαθήσει να ελέγξουμε το τι γίνεται. Λογιστικό έλεγχο στι αναπτυσσόμενε χώρε. Και έρχονται διάφοροι από οικονομική οικονομικά κέντρα από το Λονδίνο και γιατί μας λένε γιατί δεν υπάρχουν λογιστικά τα προγράμματα. Σε... Λοιπόν, προσπαθούν να μας πείσουν οι εταιρείε που κινούνται στα οικονομικά κέντρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν μπορεί να γίνει λογιστικός έλεγχος των διαφόρων προγραμμάτων που υλοποιούνται στι αναπτυσσόμενες χώρε. Δια, δια, διαβάσατε το, το βιβλίο του καθηγητού Σίλερ που λέει ότι η μείωση της σύμπραξης των ομίλων Mary Lynch, Goldman Sachs, Lehman Brothers, αυτών των συνεργασιών μειώθηκε. Όταν υπήρχε συνεργασία σύμπραξη ήταν και θέμα φήμης. Μετά όταν δεν υπήρχε θέμα προστασίας της φήμης τελικά άλλαξαν οι αξίες που περασπιζόταν. Ερώτηση για τους τρεις. Η περιορισμένη ευθύνη θα έπρεπε να η αρχή τη ε, περιορισμένη ευθύνη θα πρέπει να έρεται άμα βλέπουμε ότι ιδεολογικά κάποιο κινήθηκε λάθο. Μπορούμε αναδρομικά να αφαιρέσουμε την ε, περιορισμένη ευθύνη για να υπάρξει αντικίνητρο. Κύριε Μπέικερ, χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, κυρίως στις ΗΠΑ. Μήπως με φιλίες με το Κογκρέσο, με τέτοια μπορούν να κάνουν αυτοί που θέλουν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Στην Ευρώπη μήπως τρέχει κάτι ανάλογο. Τι έχετε να πείτε. Λοιπόν, και για τις ε, διάφορες ε, ε, εταιρείε της υπεράκτης και λοιπά που αναφέρατε. Και τις εικονικές εταιρείε. Έχουν αποδυναμωθεί οι προτάσεις του Επιτρόπου Μπαρνία για τον έλεγχο από τους μεγάλους ενεκτικούς φορείς στον κόσμο. Ε, πρέπει να υπάρχει επιτήρηση και όχι ανείχνευση τόσο πολύ. Κανονικά πρέπει να είναι λαγωνικά και τελικά είναι πούντλ αυτοί, αυτοί οι φορείς, είναι σκυλάκια. Δεν παίζουν το ρόλο που έπρεπε και οι προτάσεις του Επιτρόπου Μπαρνιέ που ήταν καλές τελικά αποδυναμώθηκαν. Ευχαριστώ κύριε Μίτσελ. Ο συνάδελφος Bill Newton Dunn έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Ε, πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Περίπλοκα, πολύ περίπλοκα τα θέματα. Έπρεπε σύντομα να παρουσιάσετε τα θέματα. Μπορούμε να έχουμε αντίγραφα των παρουσιάσεων. Ελπίζουμε να μας δώσετε, θα μας βοηθούσε να μελετήσουμε τις ε, παρουσιάσεις σας. Συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τον κύριο Μπέικερ. Μια αντιπροσωπεία θα επισκεφτεί τη Ουάσιγκτον τον επόμενο μήνα. Έχετε προτάσεις ποιο να συναντήσουμε. Παρόλο που εμείς έχουμε κάτι υπόψη μας. Δεύτερον, το FBI η ύπαρξη του FBI στη ΣΥΠΑ κάνει πραγματικά διαφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματο. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε η Ευρώπη να έχει το αντίστοιχο δικό τη FBI, δηλαδή μια διασυνοριακή αστυνομία. Για την ώρα έχουμε εκατοντάδε αστυνομικέ ε, υπηρεσίε που είναι περιορισμένε ε, συνοριακά και δεν μπορούν να δράσουν διασυνοριακά. Θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο θα έπρεπε να κάνουμε αυτό το βήμα, κατά την άποψή σα. Προ τον κύριο Μπράμλετ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε η πολιτική βούληση είναι αποφασιστική ε, σημασία. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχω κάποια ελπίδα για το μέλλον. Η δημιουργία του διαδικτύου έδωσε τη δυνατότητα στο λαό να κινηθεί. Του έδωσε εξουσία. Αυτό οδήγησε σε μεγάλη διαφάνεια. Ο οργανισμός σας κάνει κάτι. Λέτε στον κόσμο, σε όλο, τον κόσμο, πόσου εκμεταλλεύονται οι ηγέτες τους Μήπως θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τη δύναμη του λαού περισσότερο. Μήπως αυτή είναι μια διαδρομή για την επίλυση του προβλήματος. Και προς όλους τους ομίλητες. Θέλουμε κάποιες συστάσεις για δράση, για να ξέρει η Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα να κάνει. Θέλαμε συστάσεις από οτιδήποτε από εσάς. Για συγκεκριμένες δράσεις που θα έπρεπε να αναλάβουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νιούτον Ντόν. Και τώρα ο κύριος Κόρτες Λάστρα έχει το λόγο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ναι, πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω του συζητητέ και για την παρουσία του και για τι παρεμβάσει του και να του πω ότι φυσικά οποιαδήποτε ανάλυση μπορεί να γίνει μέσα σε τρία λεπτά για αυτό το θέμα θα είναι σίγουρα επιφανειακή. Θα αρχίσω από τα θετικά που είναι ίσως ότι αυτή η οικονομική κρίση, αυτή που βιώνουμε ιδίως εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοια προβλήματα και τέτοιες παγκόσμιες προκλήσεις ε, τα εντάσσει σε πρώτο επίπεδο ε, στο πολιτικό θεματολόγιο. Προκλήσεις που δεν ήταν στο πρώτο επίπεδο, στο πρώτο πλάνο, μπαίνουν τώρα σε πρώτο επίπεδο. Σίγουρα είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Επηρεάζει εκατοντάδε χιλιάδες ανθρώπου και είναι βέβαιο ότι οι νέε τεχνολογίε το λέγει ο κύριο Μπέικερ, τρεις παράδεισοι φορολογικοί υπήρχαν και τώρα είναι 60, Ίσως οι νέες τεχνολογίες συνόδευσαν παρά τη δημιουργία αυτού του φαινομένου των φορολογικών παραδείσων. Δεν συνόδευσαν όμως την ανάπτυξη νομικών ε, συμβάσεων για καταπολέμηση του εγκλήματος του οικονομικού. Κάτι που πρέπει να τονίσουμε και είναι μια πάρα πολύ σημαντική φράση, πολιτική βούληση. Ίσως δεν υπήρξε πολιτική βούληση για να ενισχυθεί η καταπολέμηση του εμπορίου όπλων, ε, του εμπορίου ε, χρημάτων, ε, της, του οργανωμένου εγκλήματος, ξεπλήματος, βρώμικρums κτλ. Δημιουργήθηκαν τεράστια ταμεία για τεράστιες περιουσίες και μπορούμε όλα να φανταστούμε πώς τροφοδοτούνται αυτά τα ταμεία. Όπως έλεγε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, με αυτή την πολιτική βούληση πρέπει να αποκτήσουμε και μεγαλύτερη ευθύνη και να δούμε ποια νομικά εργαλεία θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών με νομικά μέσα. Δεν το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και στη Λατινική Αμερική η Eurolat ε, το συζήτησε και είδαμε ότι δεν έχουμε μέσα μεταξύ χωρών για ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αφού υπάρχει τέτοια έλλειψη συντονισμού να αντιμετωπίσουμε αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα. Και το οποίο, όπως έλεγα, επηρεάζει και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Μια άλλη σκέψη, το είπε και ο κύριος Μπέικερ, είναι ζητήματα αυτά ίσως για τα οποία δεν είμαστε πάρα πολύ σκληροί από πολιτικής πλευράς. Μιλώ για τις ε, ποινές, για τις κυρώσεις, για το ξέπλυμα χρήματος, για το λαθρεμπό ναρκωτικών. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε. Πριν από λίγο καιρό, με την ε, Διεθνή Διαφάνεια, είχαμε μια συνάντηση πριν από κάποιους μήνες και είδαμε στη Βόρεια Αφρική εκατομμύρια ευρώ να εξαφανίζονται ή με ηλικιότητα ταχύτητα να μετακινούνται και να, ε, να προσπαθούν οι αρχές να παρακολουθήσουν το ίχνος τους. Πράγμα αδύνατον. Και ολοκληρώνω με αυτό. Υπάρχουν νομικά κενά. Και αυτά τα εκμεταλλεύονται αυτά τα συστήματα, οι μεγάλες τράπεζες. και τελικά εκποφελείται το χρηματοπιστωτικό τομέα ε, και όχι οι δημόσιε υπηρεσίε και βέβαια εκποφελείται έμεσα και το οργανωμένο έγκλημα και αυτά. Και ολοκληρώνω με την εξή παρατήρηση και έρχομαι στην αρχή τη ε, παρέμβασή μου. Η κρίση δημιούργησε αυτέ τι παγκόσμιε προκλήσει, μα έθεσε αντιμέτωπου με αυτέ και ε, ένα από τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η φορολογική παράδειση. Σα ρωτάω, πού ξεκινάει κανεί, πώ να ξεκινήσουμε για να καταπολεμήσουμε του φορολογικούς παραδείσου, γιατί είναι μια μάχη που πρέπει να δοθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλιώ θα είναι πολύπλοκο και δεν θα μπορέσουμε να στέψουμε, δεν μπορεί να στεφτεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρο. Κύριε Σαρτζεντίνη, το έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Σαν εισηγήτρια στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για το ξέπλυμα χρήματο και καταπολέμηση τη χρηματοδοτή τρομοκρατία, προσπαθώ να αποφασίσω. Να αποφασίσω επιπίουν ε, θέματος να προβληματιστώ. Το σχόλιο του κ. Μπέικερ με εντυπωσίασε για, το, για τη φόρα αποφυγή και το ξέπνο βρώμικου χρήματος. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι, χρησιμοποιείται η ίδια διαδρομή, η ίδια προσέγγιση, οι ίδιες οργανώσεις χρησιμοποιούν αυτή την προσέγγιση. Αν, αν αντιμετωπίσουμε το ξέπλυμα χρήματος μπορούμε να καταπολεμήσουμε και τη φόρα αποφυγή. ίσως τελικά να αντιμετωπίζεται πιο εύκολα το ξέπλυμα χρήματο από τη φοροαποφυγή. Είμαι από την Ολλανδία και το κοινοβούλιο μας είπε ότι φορολογικός παράδεισος είναι μια λέξη που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλέον, μια έκφραση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Άρα φοροαποφυγή και ξέπλυμα χρήματο. σχέση, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Δεύτερον, κάτι που δεν ανέφερε το πάνελ ακόμα. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, μετά τη θέσπιση νόμων κατά της τρομοκρατίας. Χρησιμοποιούσαν οι διάφορες δικτατορίες, ε, οι διάφορες καταπιστικές κυβερνήσεις τους νόμους αυτούς να καταπιέσουν ε, στη χώρα τους όπως οι νόμοι κατά τον ΜΚΟ στο Ζιμπάμπουε αυτό που συζητείται στην ε, Αίγυπτο για τη χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων από ξένους φορείς όπως και οργανισμοί όπως το Islamic Relief, η ε, Ισλαμική βοήθεια στην Ευρώπη που έχει πρόβλημα να δώσει χρήματα για ανθρωπιστική βοήθεια αλλού. Ε, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι με αυστηρότερη νομοθεσία εξασφαλίζουμε το ότι έχει κοινωνία των πολιτών περιθώρια να κάνει τη δουλειά που θέλει να κάνει. Αυτή είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ. Η συζήτηση θα ακολουθήσει αντίστροφη κατεύθυνση που ακολουθούν οι πορτογαλικές εταιρείε. Όχι από Πορτογαλία προς Ολλανδία, αλλά από Ολλανδία προς Πορτογαλία. Προς τη συνάδελφο Άννα Γκόμε, με άλλα λόγια. Έχετε το λόγο, Άννα. Ευχαριστώ. Κάποιοι συνάδελφοι μίλησαν για την ε, πολιτική βούληση, το είπε και ο Ρικάρντο. Αυτό που εξηγεί την έλλειψη πολιτικής ε, βούλησης είναι ότι οι πολιτικοί παγιδεύτηκαν, όχι όλοι, αλλά πολλοί, παγιδεύτηκαν από τα συμφέροντα, το οικονομικά ή, το, ή του ε, εγκλήματος ε, και στη χώρα μου, πούμε, στην Πορτογαλία, έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και έχουν υπάρξει πάρα πολύ καλές νομικές ε, δικαιολογίες που λένε ότι η παράνομη, ε, ο παράνομος πλουτισμός θα παραβίαζε την ε, θεώρηση ότι κάποιος είναι αθώος μέχρι να θεωρηθεί ένοχος. Και βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με τους φορολογικούς παραδείσους. Η φορολογική παραδείση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί και αυτοί που διαφθείρουν και αυτοί που διαφθείρονται δεν έχουν ουσιαστικά την, στην κατοχή τους ε, τα, ε, τα κλοπημαία ουσιαστικά τα χρήματα, τα κρύβουν σε, πίσω από εταιρείε ή στους φορολογικούς ε, παραδείσους. Και φορολογική παράδειση δεν υπάρχουν μόνο στα Κέιμαν, δείτε την Κύπρο. Όλοι το ξέρουν ότι η Κύπρος είναι ε, φορολογικός παράδεισος ναι, ναι. και τα καταστροφικά μέτρα που ελήφθησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και που τέλο πάντων εν μέρη διορθώθηκαν, δεν έχουν ως στόχο να σταματήσουν την Κύπρο από το να συνεχίσει να είναι φορολογικό παράδεισο για φοροδιαφεύγοντε από την Ελλάδα ή την Πορτογαλία ή για τη ρωσική μαφία. Στη ΣΥΠΑ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπέικερ. Εσείς πώς, ε, πώς μπορείτε να διαχείσετε όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται στις ΕΙΠΑ. Ε, εγώ πήγα από, με τρένο από την, από την Ουάσιγκτον στο η Νέα Υόρκη και εκεί βλέπετε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες γύρω-γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Ε, προφανώς κάποιο λόγο έχουν που είναι εκεί. Το Delaware είναι τεράστιος φορολογικός παράδεισος, όλοι το ξέρουν. Ακόμα και πολύ γνωστά και φημισμένα οικονομικά κέντρα στην, στην Ευρώπη. Οι κατοχώρες ας πούμε. Οι κατοχώρες είναι ε, φορολογικός παράδεισος για πορτογαλικές εταιρείες, το λένε σαφώς. Πάνε στην, ε, στην, ε, στην Ολλανδία για να αποφύγουν τη φορολόγηση. Όχι μόνο αυτή την φορολόγηση που δεν πληρώνουν στη στην Πορτογαλία. Είναι απλώς για να μην χρειαστεί να δηλώσουν τα χρήματα που βγάζουν στην Κίνα, στη Μοζαμβίκη, στην Αγγόλα κτλ. Ας πούμε στο Λονδίνο, το λέω συχνά, Έχουμε κάποια ε, υποβρύχια που έχουν ε, αγοραστεί από τη Γερμανία. Υπάρχει πρόβλημα δικαστικής συνεργασίας με τη Γερμανία που δεν επιτρέπει. Υπάρχουν ήδη ε, κάποιες καταδίκες, καταδίκες στην Γερμανία για, την, για τα υποβρύχια αυτά και στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί ο κύριος Μπαρόζο ήταν τότε υπεύθυνο και ο, ε, πρώην, ο πρώην Υπουργό Άμυλα στην Πορτογαλία ενώ είναι Υπουργό Εξωτερικών. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τη συνεργασία που μπορεί να υπάρξει με τις ε, Βρετανικές αρχές που θα πρέπει να ασχοληθούν. Οπότε θα ήθελα να μου το σχολιάσετε αυτό. Η Κομισιόν επίσης έχει και την οδηγία για τις αποταμιεύσεις που θα μπορεί ίσως να ε, παρακολουθεί τι γίνεται με τις αποταμιεύσεις, αλλά πόσο ξέρω αυτή η οδηγία έχει ε, μπλοκαριστεί, όχι τυχαία, από το Λουξεμβούργο και την Αυστρία. Ευχαριστώ, Άννα. Η κυρία Βάιλερ έχει το λόγο. <clears throat> ναι. Πρόεδρε, αξιότιμοι προσκεκλημένη, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν να περάσω στα δύο ερωτήματα που έχω να θέσω, θα ήθελα να πω ότι κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι το θέμα βρίσκεται πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη και ότι ε, έχουμε εμείς πλέον την ευθύνη και μπορούμε να το συνεχίσουμε. Εμείς ε, θα πρέπει να λάβουμε την ευθύνη αν θα, αν θα απλουστεύσουμε ή αν θα ενισχύσουμε την ε, νέα οδηγία του κυρίου Μπαρνιέ. Αυτή η συζήτηση ε, προφανώς αγγίζει όλες τις ε, ομάδες, οπότε στην, ε, και στις οδηγίες που αφορούν και, και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και στις υπόλοιπες επιτροπές θα πρέπει να ενισχύσουμε την παρέμβασή μας. Είναι λοιπόν η σωστή χρονική στιγμή για να γίνει αυτό για την Ευρώπη. Πέραν της Ευρώπης όμως. Το ένα ερώτημά μου είναι ότι προφανώς η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα συνδέονται πολύ στενά, αλλά τώρα στην οικονομική κρίση που έχουμε στην Ευρώπη αυτό έχει οξυνθεί ακόμη περισσότερο. Καταρχάς γιατί οι καταθέτες ψάχνουν διάφορες οάσεις αλλά και γιατί ε, το οργανωμένο έγκλημα έχει βρει καινούριου ε, δρόμους. Το ξέρουμε από τη μαφία. Ε, εξελίσσονται και δραστηριοποιούνται και σε, διαφορετικές, σε διαφορετικούς τομείς. Ερώτημα τώρα για την Αφρική. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και τις δομές της διαφθοράς και του ξεπλήματος μαύρου χρήματος στην Αφρική. Βλέπουμε ότι οι δύο μεγάλες δυνάμεις ε, ε, εξεκολουθούν να προσπαθούν ε, να διατηρήσουν ε, την ε, δεσπόλουσα θέση τους η Κίνα και η ΙΠΑ από τη μία και την άλλη πλευρά και οι δύο εμπλέκονται στον τομέα αυτό οπότε η οικονομική κρίση ρωτώ έχει οξύνει την κατάσταση στην Αφρική τι μπορεί να γίνει για να την αντιμετωπίσουμε το άλλο ερώτημά μου σχετίζεται με αυτά που είπε η κυρία Μπράμλετ για τους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι σαφέ ότι με το, με, το άτυπο τραπεζικό σύστημα είναι προφανώς πολύ δύσκολο να παρακολουθούν όλα αυτά τα χρήματα. Εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει κανείς απέναντι σε αυτό. Η βιομηχανοποίηση των μεγάλων πόλεων ε, αυξάνεται συνέχεια, οπότε οι, εργοδότες ε, πληρώνουν τους εργαζόμενούς τους μέσω τραπεζικών λογαριασμών συνέχεια αυτό γίνεται όλο και περισσότερο. Πώς μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Ας πούμε, στην Ασία πριν από πολλά χρόνια δεν, ε, δεν υπήρχαν ε, τραπεζικέ συναλλαγέ ε, με την Μιανμάρα, πούμε, για λόγους που δεν έχουν τώρα σχέση με αυτό που λέμε, αλλά υπήρξε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο ουσιαστικά προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Δημιουργήθηκαν λοιπόν κάποιες δομές για να υπάρχει σωστή τραπεζική συναλλαγή. Ε, πώς θέλετε αυτό να το επιτύχετε για την Αφρική ας πούμε ή σε βιομηχανοποιημένες χώρες. Υπάρχουν κάποια σχέδια, έχετε κάποια στρατηγική. Um Ευχαριστώ. Θα καταχαστώ το γεγονός ότι είμαι πρόεδρος για να κάνω μια ερώτηση απευθυνόμενος και εγώ προς τα μέλη του πάνελ μας εδώ. Ας φανταστούμε ότι Τρία από αυτά που προτείνατε θα συμβούν. Αναφερθήκατε στην απόδειξη. Ο κύριος Μπέικερ ήθελε να αποφύγει το φαινόμενο αυτό των εικονικών εταιριών, ε, να μπορούν να κινούνται επιχειρηματικά. Αυτό είναι απλό και πρακτικό. Και η κυρία Μπράμλετ ήθελε να θέσει δεύτερο στο, ε, να υπάρχει διάκριση μεταξύ πρωτογενού και δευτερογενούς εγκλήματος, ε, να, να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ πρωτογενού και δευτερογενού ε, αδικήματος και να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Το ερώτημά μου είναι τι θα συμβεί από τώρα και στο εξή. Πώς μπορούμε την μαύρη οικονομία, ποιο τμήμα της μπορούμε να αποκαλύψουμε και να το εντάξουμε στην κανονική οικονομία Και είχαμε και την ερώτηση συναδέλφου Γκόμε, ε, που μάλλον θα μπορούσε να απαντηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οδηγία για τι αποταμιεύσει κλπ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο να σχολιάσει. Άρα να δώσουμε το λόγο ξανά στα μέλη του πάνελ για να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις. Πρέπει στις 10.45 να ολοκληρώσουμε τις εργασίες. Παρακαλώ είστε σύντομοι. Ο καθένας ένα πεντάλεπτο να ακολουθήσουμε την ίδια σειρά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις. Ευρύ το φάσμα των ερωτήσεων που ετέθησαν. Δεν μπορούσα να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Πάμε στην πρώτη ερώτηση, λαμβάνοντας υπόψη και το τέταρτο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αν εφαρμοζόταν σωστά τα μέτρα, δηλαδή ποινικοποίηση του ανεξήγητου πλούτου ε, να ενταχθεί σε νομοθεσία και αν διωχθεί το φαινόμενο αποτελεσματικά, πιστεύω ότι θα είχε σημαντική επίδραση όσον αφορά στις διεφθαρμένες πρακτικές που ακολουθούνται στη δημόσια διοίκηση. Από ό,τι είδαμε στο Χονγκ Κονγκ, ίσως δεν είναι ενδεικτικό για το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, χρησιμοποιήθηκε αυτή η προσέγγιση για να σπάσει ο κύκλος ε, της διαφθοράς. Όταν δεν υπήρχε από την αρχή βέβαια κάτι εμφανές, εμφανές στοιχείο ότι υπάρχει ε, διαφθορά. Εκεί που εργαζόμουν εγώ στην Ανατολική Ευρώπη, μια προσέγγιση ε, παρόμοια θα είχε χαμηλότερα, μικρότερα αποτελέσματα, χρήσιμα αποτελέσματα, αλλά πιο μέτρια. Γιατί? Το θέμα επιβολής του νόμου. υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά αυτό η ανεξαρτησία ε, της δίωξης των διοκτικών αρχών και η ανεξαρτησία των δικαστηρίων είναι κάτι που είναι προβληματικό. Ε, θα πρέπει τελικά να υπάρχει σωστή επαφή διοκτικών αρχών. Με, κυρίως στις μικρές χώρες υπάρχει το πρόβλημα. Υπάρχει ε, αλληλοκάλυψη και δεν υπάρχει πληροφόρηση και ενημέρωση των διοκτικών αρχών. και αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα με κατάχρηση εξουσίας ο ΣΥΠΗΝ ή αμέλεια πλημελής εκτέλεση καθηκόντων που προσπαθούν να... Οι αρχές να χρησιμοποιήσουν αυτές τις προσεγγίσεις και δεν καλύπτεται το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό. Ο κύριος Μίτσελ έθεσε ένα ερώτημα. Η Δημοκρατία της Ιρλανδίας με το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κάποια κοινή προσέγγιση. Υπάρχει υπηρεσία για παράνομα, παράνομες και υπάρχει και η δυνατότητα αντιστροφή του βάρου τη απόδειξη. Πρέπει ο ύποπτο να εξηγήσει στην Ιρλανδία το πόθεν Έχουμε τρία επίπεδα στη Βρετανία. Έχουμε ποινική δίωξη. Βλέπει κανεί ποια είναι τα στοιχεία ενεργητικού του καταδικασμένου που αντιστοιχούν στο εγ... θεωρούνται ότι είναι αντίστοιχα στο έγκλημα και στον τρόπο διαβίωσης. Αν καταδικαστεί για κάποιο επίπεδο εγκλήματος μπορείς να πάρεις αναδρομικά περιουσιακά του στοιχεία, διότι υποθέτει ότι είναι προϊόντα του παρανόμου τρόπου ζωή του και εκείνο ή εκείνη πρέπει να αποδείξει ενισχύει αυτό κάτι τέτοιο. Αν δεν λειτουργήσει ποινική προσέγγιση, υπάρχει μη ποινική ή η αστική, η αστική κατάσχεση. Το κράτο πρέπει να αποδείξει με στάθμιση πιθανότητων ότι ο τρόπο ζωή και ο πλούτο του ατόμου ε, είναι προϊόν εγκλήματο. Και αν δεν λειτουργήσει και αυτό υπάρχει τρίτη προσέγγιση το φορολογικό σύστημα. Ολιστική προσέγγιση για τα προϊόντα εγκλήματος χρειάζεται. Σχόλιο. Εν είδη πρόκλησης. Είδα το σχέδιο έκθεσης. Ασχολούμαι με τα ποινικά θέματα ίδιος. Είμαι εισαγγελεύς. Δεν μιλώ εκ μέρους της εισαγγελικής αρχής. Μιλώ προσωπικά έχω την εξή εντύπωση. Σε μια χώρα που εφαρμόζεται ο νόμος, πάντα εμείς θα είμαστε πίσω από το οργανωμένο έγκλημα. Η μόνοι ειδικοί όσον αφορά το ξέπνο χρήματο είναι οι οργανωμένοι εγκληματίε. Πάντα βρίσκουν τρόπου να ξεφεύγουν. Είναι επιδέξι, είναι αποτελεσματική. Είναι ευάλωτοι μόνο από δύο πλευρέ. Πρώτον, σχετικά λίγοι άνθρωποι αναμειγνύονται με το όλο σύστημα. Δεύτερο στοιχείο ευαλωτότητας. Προσπαθούν να μετακινήσουν πολύ μεγάλα ποσά σε ρευστό από χώρα σε χώρα στον κόσμο. Ίσως να υπάρχουν διαφωνίες με τα δύο αυτά σημεία που ανέφερα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι μόνο πιάνουμε περιορισμένο αριθμό εγκληματιών. Καλύπτουμε περιορισμένο ποσοστό αυτών των παρανόμων ποσών, το 10%. Κάποιε χώρε τα καταφέρουν κάπω καλύτερα. Γιατί είμαστε χώρε όπου εφαρμόζεται ο νόμο. Τι γίνεται με το 90%. Αυτό δεν το καλύπτουν οι επιτροπές, έτσι πιστεύω. Καταλαβαίνω γιατί. Έχετε δυνατότητα να συλλέξετε στοιχεία από διάφορες πηγές. Μιλάμε για τη δημιουργία δυναμικού εναρμόνιση νομοθεσίας, επίδυση από δικαιοδοσία σε και δικαιοδοσία, ευρωπαϊκό FBI, σε κάποια περίπτωση αναφέρθηκε, ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Όμως, τι κάνουμε για να εργαστούμε στο μη ποινικό επίπεδο. Τι κάνουμε για την πρόληψη διάπραξη των αδικημάτων. Και κάτι σημαντικό. Τι κάνουμε για να δημιουργήσουμε προβλήματα, αν δεν μπορούμε να καταδικάσουμε για να τους εμποδίσουμε τις ε, ροές των χρημάτων. Το ξέπλυμα χρήματος και η σχετική νομοθεσία περιέχει ισχυρότατους μηχανισμούς ελεγκτικούς. Οι, οι, ελε, φορεί πρέπει ε, αντιπροσωπείς αυτοκινήτων, παραδείγματος χάρη, διάφοροι φορείς θα πρέπει να αναφέρουν το τι γίνεται. Ε, οι μεσίτες ακινήτων περνάνε δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως στο Λονδίνο δισεκατομμύρια ευρώ περνούν τα χέρια τους δεν υποβάλλουν εκθέσεις, δεν αναφέρουν σε κανέναν. Ίσως εκεί έγκυται η, η λύση. Ευφυής παρεμπόδιση ε, ροής αυτών των χρημάτων είναι το κλειδί. Αν δεν μπορείς να διώξεις, χρησιμοποίησε ευφυείς πηγές να βρεις ποιοι κάνουν το ξέπλυμα του χρήματος. Και μετά πήγαινε να τους ελέγξεις, να ελέγξεις τα στηριότητες τους. Αυτό είναι νόμιμο. Είμαι ένοχος. Συγγνώμη. Ε, ξεπέρασα το χρόνο μου, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν ε, μπόρεσα να αντισταθώ στον πειρασμό να ξεφύγω λίγο από το όριο. Απαλλάσσεστε, κύριε Βινίνγκ, ο κύριος Μπέικερ. Um, um, uh, Προς το δικό σας ερώτημα, θέλω να διευκρινίσω ότι εγώ είμαι υπέρ του συστήματος της ελευθερής αγοράς. 35 χρόνια ήμουν σε επιχειρήσεις και ασχολούμουν με τον αψόμενο κόσμο και μετά πήγα σε μια ε, ομάδα σκέψης. Βέβαια όλα αυτά τα ελεύθερα πρέπει να είναι και νόμιμα. Αυτό είναι το, το ζήτημα. Για τον κύριο Μίτσελ. Φυσικά και μπορούν οι εταιρείε ε, ε, σε μια βάση project ανά project να λογοδοτούν. Το προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Ε, μπορούν να υπάρξουν βέβαια παράπονα, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί. και προβλήματα υπήρξαν όταν έπρεπε να λογοδοτούν επιχειρήσεις χώρα προς χώρα. Παρ' όλα αυτά γίνεται. Πολύ σωστά Μιλήσατε για τις εταιρείε περιορισμένη ευθύνη. Πραγματικά ουσιαστικά αυτό το οποίο σημαίνει όρος περιορισμένη ευθύνη το έχουμε κάπως διαστρεβλώσει γιατί κάναμε να περιλαμβάνει και την έννοια της εμπιστευτικότητας. Δεν ήταν όμως αυτή η έννοια της περισμένης ευθύνης πριν από 200 χρόνια και ότι και σήμερα θα έπρεπε να είναι να μπαίνει μέσα η εμπιστευτικότητα, το απόρριτο, η μυστική ε, δραστηριότητα. Επίσης, πολύ σωστά είπατε για τους ελεγκτές. Οι ελεγκτές μπορούν να δουν παραδείγματα φοροδιαφυγής στους ελεγμένους λογαριασμούς ε, συνεχώς, αλλά δεν υποχρεούνται να το σημειώσουν στους εκκριμένους λογαριασμούς αυτό. Σε πολλές αντισόμενες χώρες ε, συστήσαμε να γίνει μια απέτηση. Αν δηλαδή μια εταιρεία ελέγχου δει τέτοια ε, στοιχεία, να απαιτείται να το σημειώσει αυτό ο λογαριασμό για τον κύριο τον Ντάν. Μπορούμε να συζητήσουμε ε, για αυτή την αντιπροσωπεία που θα τη συστήση, Είπατε κατά πόσο πρέπει να δημιουργηθεί μια διασυνοριακή αστυνομία κάνω ότι δεν άκουσα, γιατί δεν έχω να σας απαντήσω. Παρακάμπτω αυτό το ερώτημα. Ε, περνάω τώρα στο άλλο σας ερώτημα για τις συστάσεις ε, το δικό σας σχόλιο, κύριε Λάστρα, και το σχόλιο της κυρίας Γκόμες, ιδίως ό,τι αφορά τους φορολογικούς παραδείσους. Πώς μπορούμε να περιορίσουμε ε, τις δραστηριότητες, όχι να επιτεθούμε στην κυριαρχία του στο δικαίωμα να υπάρχουν αυτοί οι φορολογικοί παράδεισοι, δεν μπορούμε να του το απαγορεύσουμε να υπάρχουν, αλλά έχουμε δύο θέματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Το απόρριτο, τη μυστικότητα μάλλον και την απόκρυψη των εταιρικών κερδών. Εάν την ε, ιδιοκτησία τους την αφαιρέσουμε και ζητηθεί να υπάρχει αναφορά reporting ανά project, ουσιαστικά κόβουμε τα πόδια στους περισσότερους φορολογικούς παραδείσους δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης. και σε ό,τι τον beneficial owners. Δηλαδή δεν θα έχουμε πλέον μυστικές δικαιοδοσίες, φορολογική παράδειση. Η χρήση τους θα μπορούσε σχεδόν να εξελιχθεί. Αναφορά χώρα προς χώρα και υποφελής ε, ιδιοκτησία αν υπάρχουν τώρα περιθώρια μόνο για τις ΜΚΟ. Είναι πρόβλημα. Το βλέπουμε στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες. Είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Επίσης πρέπει να προσέξουμε και την ε, κακή χρήση των ΜΚΟ. για τον Delaware και όλα αυτά που είπατε έχουμε και καλυμμένες εταιρείε της ΕΠΑ πολύ περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και αυτό διότι στις ΗΠΑ στο επίπεδο πολιτείας ε, υπάρχει ευθύνη. Δεν υπάρχει εταιρική ε, εταιρεία. Με, συγγνώμη, ομοσπονδιακή εταιρεία. Είναι σε επίπεδο πολιτείας. Τώρα έχουμε πάνω από 40 πολιτείες της ΕΥΠΑ που επιτρέπουν το σχηματισμό εταιριών από συγκεκριμένα άτομα που μόνο αυτά γνωρίζουν τα φυσικά πρόσωπα. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει τις διεκτικές αρχές, τις αρχές επιβολής του νόμου. Και πρέπει να αλλάξει. Σας είχα πει ότι η ηγεσία στα ζητήματα αυτά μετατοπίζεται προς την Ευρώπη και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης που μιλήσατε για την Αφρική. Έζησα 15 χρόνια εκεί και έτσι με συνδέουν πολύ βαθιά αισθήματα έκτοτε με αυτή την ε, Ήπειρο. μέσω της Οικονομικής Επιτροπής για την Αφρική, του ΟΗΕ, που έχει ένα μια επιτροπή με πρώτα τον πρώην πρόεδρο της Νοτιοαφρικής Μπέκη. Ελέγχει τη μεταφορά ε, οικονομικών ροών. Κάναμε και μια έκθεση για την Αφρική πριν από κάποιες χώρες, κάποια, κάποια χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν τις παράνομες ροές από Αφρική προς άλλες χώρες. Αυτό το κάνουμε μαζί με την, ε, τράπεζα, την Αναπτυξιακή Αφρικανική Τράπεζα. Και θα έχουμε τα πορίσματα στη δημοσιότητα πολύ σύντομα. Τι γίνεται με αυτές οι ιονίκονικές εταιρείε. Εάν τις βγάλουμε εκτός δραστηριότητας, τις ποινικέ, εγκληματικέ, αυτές δεν θα περάσουν στην ε, κανονική οικονομία, στην νόμιμη οικονομία Όποιες είναι στι παρυφές όμως ναι, θα μπουν στην νομιμή οικονομία. Και δεν νομίζω ότι αν αυτές τις ε, εταιρείε τις βγάλουμε από την δραστηριότητα θα δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα. Ναι, αυτό που είπατε κύριε Μίτσελ επίση, ε, η αναγνώριση των εταιριών ως προσώπων ήταν κάτι τρομερό, γιατί εταιρείε τη είπα, μπορούν να χρηματοδοτούν πολιτικά, πολιτικές εκστρατείες από τη στιγμή που αποφασίστηκε ότι η εταιρεία είναι πρόσωπο στο Μέριλαντ, μια εταιρεία, ε, υπέβαλε ε, υποψηφιότητα για το αξίωμα του πρόεδρου. Εντάξει, φυσικά αυτό δεν είναι δυνατόν, αλλά σας ε, δείχνω το γέλιο της όλης υπόθεσης και της νομοθεσίας αυτής. Η χρηματοδότηση λοιπόν ε, των εκλογών από εταιρείε είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλέ περιπτώσει πολιτικοί εξαγοράστηκαν ουσιαστικά λόγω αυτού του μηχανισμού χρηματοδότηση των εκλογών. Ε, τότε θα θέλουν, λέει ο κύριο Σταβάρη, ε, οι εταιρείε, αν είναι πρόσωπα, να παντρεύονται και να κάνουν και παιδιά. Ε, η, η, κυρία του πάνελ τώρα. Ναι, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη για να μην ξεπεράσω το χρόνο που μου διαθέσατε γιατί είπατε ότι πρέπει παρατέταρτο να έχουμε ολοκληρώσει. Στον κύριο Βαντεμίρ θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τη σταθερότητα. Ε, είπατε ότι εστιάζεται πιο πολύ στην καταπολέμηση του λαθρομπόριου ναρκωτικών. Η Επιτροπή ε, για την καταπολέμηση των ναρκωτικών που συζητήσαμε στο UNODC συσχετίστηκε το θέμα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και του ξεπλήματος χρήματος που πρέπει να είναι και μια ενεργό συνιστόσα στην καταπολέμηση του λαθρομπορίου ναρκωτικών. Στην πλευρά του ΟΗΕ μπορούμε λοιπόν ήδη να κάνουμε αυτή τη ε, διασύνδεση. Ίσως θα πρέπει να γίνει και ό,τι αφορά την ενίσχυση περιφερειακή συνεργασία. Υπάρχουν πλατφόρμε για τη Λατινική Αμερική και σε ό,τι αφορά ε, την ανάκτηση δίμευση περιουσιακών στοιχείων. Έχουμε ε, κάποια άτυπα δίκτυα τα οποία βασίζονται σε ένα δίκτυο που έχουμε τώρα με γραμματεία στη Europol. 65 μέλη και παρατηρητές περιλαμβάνει. Ξεκίνησε με τα κράτη της Ένωσης και επεκτείνεται και το μοντέλο χρησιμοποιείται και στην Νότια Αφρική. Έχουμε το RAG που θα συνδεθεί με την GAF και έχουμε και την ARINZA. Επομένως, οικονομικοί ανακριτές ή εισαγγελείς συνεργάζονται, ανταλλάσσουν πληροφορίες και άλλοι επιμορφώνονται, εκπαιδεύονται για την εντοπισμό και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να διευκολυνθεί συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών σε αυτούς τους κλάδους. Ό,τι αφορά τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, την ε, κατάχρηση, ε, την εκμετάλλευση που παρατηρείται. Πράγματι κάποια αγαθαργή ιδρύματα μπορεί να τα εκμεταλλεύονται κάποιοι τρομοκράτες, τελικά να χρηματοδοτούν τρομοκρατικές δραστηριότητες ή να συμμετέχουν στο ξέπλυμα χρήματος. Τελικά το θέμα είναι αν θα υπάρχουν νόμοι και εποπτικές αρχές από τα κράτη για να παρακολουθούν τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, και αν μπορούν να τα ε, να επιβάλλουν κυρώσει αν διαπιστώσουν παράνομη συμπεριφορά. Για την πολιτική βούληση ακούστηκαν πολλά πράγματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σε ανώτατο επίπεδο του ΟΗΕ, οι αξιωματούχοι μαζί με του κυβερνητικού αξιωματούχου ε, ε, βλέπουν το ζήτημα αυτό τη πολιτική βούληση το ΦΑΤΦ, η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, επιβάλλει κυρώσεις σε που δεν ε, συμμορφώνονται τους, ε, με τους κανόνες της. Σας μίλησα για αυτό το μαύρο κατάλογο, το blacklist, αλλά έχουμε και καθεστώς ε, κυρώσεων από αυτή την δικαιομάδα. Ομάδα. Άρα μέτρα υπάρχουν, κάποια μέτρα. Βέβαια, οι κυβερνήσει είναι αυτέ που είναι υπεύθυνε να ασκήσουν πιέσει η μία προ την άλλη για να τηρούν διεθνή πρότυπα, διεθνού κανόνε και για να ασκούν την πολιτική βούληση για την καταπολέμηση ε, των παράνομων χρηματοοικονομικών και του ξεπλήματος χρήματος ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών να μπορεί να λειτουργεί ε, σε επίπεδο και σε πλαίσιο πιο μεγάλων περιορισμών του ξεπλήματος χρήματος. Το γνωρίζουμε σε επίπεδο ΟΗΕ στην ε, διεύθυνση που παρακολουθεί και την εκτέλεση ψήφου του 1973 βλέπουμε και θέλουμε να προωθήσουμε την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή της ε, νομοθεσίας ε, σε όλο το σύστημα του Υπάρχουν ειδικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ενεργά εργάζονται σε αυτόν τον τομέα και υπάρχει και ένα παγκόσμιο πρόγραμμα σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη σε περιφερειακό επίπεδο, εκεί επισημαίνουμε την κατάχρηση και την εκμετάλλευση ΜΚΟ και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Θέλω επίσης να επισώ την προσοχή σας σε ένα μοντέλο που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Charity Commission of England and Wales. Είναι καλή πρακτική, είναι σχεδόν κυβερνητικός ο φορέας αυτός και σε πολλές πρακτικές του ΟΗΕ και στο έργο μας το επισημαίνουμε. Αυτή η πρακτική είναι θετική αυτού του οργανισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουαλία. Για τους λογαριασμούς που είπατε, πράγματι είναι δύσκολο να ρυθμιστούν πολλά πράγματα. Ένα σύστημα που χρησιμοποιείται στη Σενεγάλ και την Κάμπια, για παράδειγμα, το οποίο στηρίζεται από την Total ε, η οποία ενθαρρύνει ε, τους ε, υπαλλήλου της να χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα εμβασμάτων. Το θέμα είναι να καταγράφεται ε, ο κόσμος που το χρησιμοποιεί. Είναι ίσως απλό να τους βάζουμε να δείχνουν ταυτότητα και οι τράπεζες να υποχρεούνται να αναφέρουν. Δεν είναι τόσο δύσκολο, απλά οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με τους διαφόρους θεσμούς, να διαδοθούν πληροφορίες αυτές συστηματικά, να εκπαιδευτούν ε, οι οικονομικοί ελεγκτές, ε, οι άνθρωποι που έχουν ε, ευθύνη στον τομέα του reporting. Εμείς τονίζουμε ως γραφείο του ΟΗΕ τα σχετικά. Και εδώ ολοκληρώνω. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ε, φτάσαμε στο τέλος μια πολύ πλούσια πολύ ε, Έχουμε τον κύριο Μαρτίνες και τον κύριο Νιούτον Ντάν, οι οποίοι θα αναλάβουν ε, να προεδρεύσουν του επόμενου πάνελ. Ζητώ λοιπόν την ανοχή τους για λίγα λεπτά για να δώσουμε τον λόγο στη συμπρόεδρο, στην Εύα Ζολή, να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εν ονόμα της Επιτροπής Ανάπτυξης θέλω να πω ότι κανένα άλλο θέμα δεν είναι τόσο σημαντικό για την μοίρα των αναπτυσσομένων χωρών όσο το θέμα των φορολογικών παραδείσων και η καταπολέμηση του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. Ε, πώς να σας το πω τώρα. Είμαστε σε μια κατάσταση ε, κρίσιμη θα έλεγα, προφανώς. Έχουμε φυλακιστεί από τα συστήματα που δημιουργήσαμε. Βλέπουμε την υποκρισία Βλέπουμε την Κύπρο. Τι είναι η Κύπρος. Τι είναι το φορολογικό καθεστώς της Ολλανδίας. Είναι υποκριτικό αυτό που κάνουμε. Βλέπουμε το εμπόριο του ε, ρωσικού χρήματος που είναι κλοπή ε, των χρημάτων των Ρώσων πολιτών. Το βλέπουμε που συμβαίνει. Και σήμερα που καταραίει το σύστημα ε, θα θέλαμε να μην ενοχλήσουμε πολύ τους Ρώσους ώστε να συνεχιστεί η ροή του παρανόμου χρήματος. Βλέπουμε ότι το φορολογικό καθεστώς το Ολλανδικό που δημιουργεί τόσο μεγάλα προβλήματα στι αναπτυσσόμενε χώρες δημιουργήθηκε για να επιτρέπει ακριβώς αυτό, να μην πληρώνονται οι φόροι στις χώρες που έχουν τους πόρους για να αυξηθεί το μερίδιο, το μέρισμα των μετόχων σε αναπτυγμένες χώρες. Και το ίδιο ισχύει και για το ΣΥΤΙ. Η ώρα της αλήθεια ήρθε. Η ευθύνη είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε τώρα να πάρουμε στα σοβαρά αυτά τα ζητήματα, τα ζητήματα αυτά που έβλαψαν τόσες χώρες. Και επιτέλους να δημιουργήσουμε ένα ρυθμιστικό σύστημα σοβαρό. Ήτι την υποχρέωση ενημέρωσης χώρα με χώρα. και να υπάρχει ενημέρωση ε, καταθέσεων σε ξένη χώρα. Να αναφερθώ και στο Αφγανιστάν, που είναι θύμα διαφθοράς και ξεπλήματος. Δεν υπάρχει πρόβλημα έλλειψης γνώσης. Είναι ενοχή ε, βούληση ε, του να πλουτίσουν εις βάρος του πληθυσμού από την υπόθεση Καμπούλ Bank. Ε, βλέπετε την έκθεση που υπάρχει στην ιστοσελίδα μου. Ο Αυγα... Οι Αυγανοί ζήτησαν τη συνεργασία των κέντρων των offshore, ζήτησαν από το Ντουμπάι συνεργασία για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Ζήτησαν από ευρωπαϊκές χώρες, ζήτησαν τη Γαλλία συνεργασία. Δεν υπήρξε απάντηση. Και αυτό δεν οφείλεται σε έλλειψη γνώσης. Το ότι δεν συνεργάζονται αυτά τα υπερπόδια κέντρα, τα, τα offshore centers. Ε, αυτά τα κάνει, αυτό τα κάνει να λειτουργούν. Δεν πρέπει να δεχόμαστε πλέον αυτό το άδικο σύστημα. Τα συστήματα αυτά που σχεδιάστηκαν για να πλουτίσουν κάποιοι εις βάρος κάποιων άλλων. Ευχαριστώ Εύα. Και τώρα ο κύριος Μαρτίνες και ο κύριος Νιούτον Ντάν έχουν το λόγο για να... και θα διευθύνουν τη συζήτηση για το δεύτερο μέρος του... των εργασιών μας. Ευχαριστώ.

Sí. señoras y και κύριοι, καλημέρα σας. Θα συνεχίσουμε την ε, ακρόασή μας για σήμερα το πρωί. Χαίρομαι πάρα πολύ πως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, λαμβάνω το λόγο βέβαια, είμαι και μέλος Επιτρόπης Ανάπτυξης, στην οποία πολύ καιρό εργαζόμαστε για όλα αυτά τα θέματα. Θα είμαι λοιπόν συμπροεδρεύων αυτή της δεύτερης, του, του δεύτερου πάνελ σε ό,τι αφορά τη διαφθορά των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Όσου, μιλάμε για όσους έχουν πολιτικό αξίωμα. Μπορεί να μην είμαστε όλοι υπάλληλοι, αλλά λειτουργοί είμαστε. Το λέω αυτό γιατί στα γαλλικά και στα ισπανικά δεν είναι ακριβώς ο ίδιος όρος. Συμπροεδρεύει και ο κύριος Μπίλ Νιούτον Ντάν που υπήρξε κοσμήτορα για πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο, άρα ήταν ε, μεταξύ άλλων ε, αρμόδιος και για τα θέματα της διαφάνειας. Της διάβγεια, αν θέλετε, όλων των δραστηριοτήτων και δι ε, των εμπορικών δραστηριοτήτων που δεξάγονται εδώ στο Κοινοβούλιο. Στο Προεδρείο Έχουμε τον κύριο Σαϊντ Πάρτο, διευθυντή έρευνας στην Afghanistan Public Policy Research Organization, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μία μελέτη για τη διαφθορά στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοικοδόμησης του Αφγανιστάν. Είναι επίσης εδώ ο κύριος Σοφίρ Ντρόντι από το Wildlife Law Enforcement, θα μας μιλήσει για τις διασυνδέσεις μεταξύ διαφθοράς οργανωμένου εγκλήματος στις χώρες ε, ανάπτυξη και συγκεκριμένα θα μας μιλήσει για τις ε, εγκληματικές πρακτικές κατά της άγριας και προστατευόμενης πανίδας και έχουμε και την κυρία Πέτρα Κνόιερ, της Όλα, διευθύντρια συγγνώμη της Όλαφ, που θα μας μιλήσει για το ευρωπαϊκό πλαίσιο καταπολέμησης και πρόληψης της διαφθοράς αναπτυσσόμενες χώρες. Ήθελα να κάνω τέσσερις ε, δηλώσεις κηρύσσοντας έτσι την έναρξη και της δεύτερης αυτής, ε, του δεύτερου σκέλους της ακρόασης. Θέλω να συγχαρώ την συνάδελφό μου Εύα Ζολή γιατί ήταν πάρα πολύ εύστοχη η διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Πρώτη δήλωση. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι πολυσχηδής και παγκοσμιοποιημένη διαφθορά. Νομίζω ότι ετέθη και δεν χωρεί αμφισβήτηση και από το πρώτο πάνελ κυρία Ζολή, κλείνοντας το πρώτο στρογγυλό τραπέζι, είπε και τόνισε ότι η διαφθορά ουσιαστικά είναι θεσμοθετημένη λόγω των φορολογικών παραδείσων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν μπορέσουμε να προβούμε σε μια δημοσιονομική ένωση στις χώρες μας, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Αν δεν υπάρχει δημοσιονομική ένωση, δεν θα έχουμε δυνατότητα να λύσουμε το πρόβλημα των φορολογικών παραδείσων. Δεύτερη δήλωση, που σχετίζεται βέβαια σαφώς και με την πρώτη. Δεν θα υπήρχε διαφθορά, είναι προφανές αυτό, δεν θα υπήρχαν και διεφθαρμένοι αν δεν υπήρχαν διαφθορείς. Οι διαφθορείς δεν είναι σαν αναψώμενες χώρες, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μεταξύ μας. Κινούνται ανάμεσά μας, κυρίως. Υπάρχουν διαφθορείς πέμπτης κατηγορίας ε, και σαν αναψώμενες χώρες, που ουσιαστικά όμως παραλαμβάνουν ε, τη διαφθορά που ε, πηγάζει εδώ από εμάς στις ε, αναπτυγμένες χώρες. Και εδώ πρέπει να αναζητήσουμε τις ρίζες της διαφθοράς για να την αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα. Επειδή ακριβώ οι διαφθορή είναι μεταξύ ημών, ίσω και αυτός είναι ο λόγο που μεταξύ μα δεν καταφέραμε να βρούμε μηχανισμούς διαφάνεια, μηχανισμούς ε, άμυνα και προστασία ε, από την διαφθορά. Τρίτη παρατήρηση. Είναι καταστροφικές οι επιπτώσεις ε, της διαφοράς στην ανάπτυξη. Μου ετοίμασαν ε, ένα προσχέδιο από την Γραμματεία της Επιτροπής Ανάπτυξης και υπάρχουν ε, κάποια συγκεκριμένα σημεία που περιγράφουν πολύ συγκεκριμένα την κατάσταση θα τα πούν και τα μέλη του πάνελ. Είναι καταστροφικές οι επιπτώσεις, αλλά γενικά είναι μεν καταστροφική, ακόμα πιο καταστροφική όμως είναι ειδικά για την ανάπτυξη διαφθορά. Για το Αφγανιστάν θα ακούσουμε, είπε ορισμένα πράγματα ήδη κυρία Ζόλη. στο Επιτροπή Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου είχαμε και σημείο στη Μεσιά Διάταξη. 900 εκατομμύρια ευρώ ως διαμαγιάς εξαφανίστηκαν. Και ποιος τα πήρε, ο αδερφός του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος. Και πού βρίσκονται τώρα. Άντε να βρεις. Πού πήγαν αυτά τα 900 εκατομμύρια. Δεν δίνεται η πληροφορία. Ποιος θα κρυφθεί, ποιος θα διωχθεί. για αυτή τη λαθροχειρία. Και πώς θα αποτρέψουμε αυτό το φαινόμενο να επαναληφθεί και να ξαναεπαναληφθεί. Σκανδαλώδη αυτή η κατάσταση, το είπε και η κυρία Ζολή χθε. Αν δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε αντίστοιχα κρούσματα. Ο κύριος Σπάρτο θα μας παρουσιάσει τη μελέτη αυτή που ελπίζω να μας κάνει και να κινητοποιηθούμε ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Τελευταία, τέταρτη παρατήρησή μου. Να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν θέλω να κάνω τη διαφήμιση σε κανέναν οργανισμό και δεν θα αναφέρω, δηλαδή δεν κατονομάσω κανέναν οργανισμό και είμαι και αρκετά επιφυλακτικός και ε, απέναντι σε όλα αυτά. Αν δούμε όμως τι γίνεται σε χώρες με μεγάλη διαφθορά, Πραγματικά μας σηκώνει τη τρίχα άμα δούμε τα ποσά. Γιατί άκρος διεφθαρμένες είναι χώρες με τις οποίες έχουμε σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν αναπτυξιακή βοήθεια, αναπτυξιακή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτος δωρητή στον κόσμο και βέβαια ε, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη. Αν δει λοιπόν κανεί την κατάταξη, αν δει την ταξινόμηση των χωρών με τη μεγάλη και την πιο γενικευμένη διαφορά, ε, βλέπει ότι από τις χώρες ΑΚΕ, οι εταίροι μας, με εξαίρεση την Καραϊβική, που είναι σε μια δεύτερη ή τρίτη στήλη, οι χώρε της Αφρικής με τις οποίες εμείς συνεργαζόμαστε είναι στην κορυφή. Στην πρώτη λίστα δεν υπάρχει κανένα, 25, στη δεύτερη ναι. Μία χώρα και στην τελευταία, την τρίτη, όπου υπάρχει ενδυμική διαφθορά, εκεί βλέπουμε να είναι η εταίροι δική μας. Θέλω να ακούσουμε την Κομισιόν κάποια στιγμή. Να μας πει κάποια στιγμή Κομισιόν πώς είναι δυνατόν οι δικοί μας εταίροι στην ε, διαδικασία αυτή της αναπτυξικής συνεργασίας να καταγγέλλονται μεταξύ χωρών με πάρα πολύ μεγάλη διαφθορά. Πραγματικά αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και να μας απασχολήσει τα μάλα. Αυτά ήθελα να πω εν είδη εισαγωγή για αυτό το στρογγυλό τραπέζι. Υπόθηκαν πολλά και σημαντικά πράγματα στο πρώτο στρογγυλό τραπέζι και με βάση αυτά, με αφετηρία τα όσα υπόθηκαν στην προηγούμενη συνεδρία, θα συζητήσουμε εμείς τώρα. Πριν δώσω όμως το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας, θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου, τον κύριο Νιτον Ντάν για να παρουσιάσει και αυτός το ζήτημα για το οποίο σήμερα θα συζητήσουμε. Uh, thank you, Mr. President. Very briefly, because... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα, γιατί περνάει ο χρόνος και ήδη έχουμε αργήσει, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον το πρώτο πάνελ. Η ουσία αυτή τη συνεδρίαση και τη δουλειά που κάνουν και η Επιτροπή Ανάπτυξη και η Επιτροπή Κριν και χαίρομαι που είμαι μέλο και στι δύο, είναι ότι ο απλός ε, κόσμος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον αναπτυσσόμενο κόσμο υποφέρει λόγω ακριβώς της δωροδοκίας και της διαφθοράς όσων βρίσκονται στην εξουσία. Όλοι υποφέρουν και αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία το εκμεταλλεύονται. Αυτό βεβαίως ίσχυε πάντα. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι το θέμα αυτό επιτέλους ε, μπαίνει σε, στις πρώτες θέσεις των, ε, της ημερής διάταξης και αρχίζουμε να επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Όσο λοιπόν γίνεται όλο και πιο σημαντικό, αυτό που ακολουθεί είναι να αναλάβουμε δράση. Ή θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Κινούμαστε λοιπόν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και παρά το ότι η δουλειά που κάνουμε σε αυτή την ακρόαση σήμερα δεν έχει να κάνει με την ομοθετική δουλειά, έχει να κάνει με την επισημοποίηση της πολιτικής βούλησης στην Ευρώπη. Τι θέλουμε. Αν μπορέσουμε να έχουμε, να δώσουμε ένα αυστηρό μήνυμα, τότε θα ακολουθήσουν και οι δράσεις. Όλοι λοιπόν εδώ μέσα στην αίθουσα εμπλέκονται σε αυτό. Όλοι μπορούν να βοηθήσουν καθώς επίσης και όσοι μας παρακολουθούν από το ίντερνετ μπορούν να συμβάλλουν ε, στην αντιμετώπιση της διαφθοράς για να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο, μια καλύτερη ζωή για όλους όσους δεν εμπλέκονται με τη διαφθορά. Περνάει λοιπόν ο χρόνος πρόεδρε, οπότε σας ξαναδίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Μπιλ. Να δώσουμε λοιπόν τώρα κατευθείαν το λόγο σε πυρογνώμονε μας. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσει ο κύριο Πάρτο. Έχετε κύριε Πάρτο 15 λεπτά στη διάθεσή σας για μια παρέμβαση την οποία περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Uh, thank you very much for um, us here. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την υποδοχή σας. Ελπίζω να μην απογοητευτείτε μετά από τα όλα καλά υπόθηκαν για την παρουσίασή μου. Υπάρχουν κάποιες διαφάνειες PDF, μπορείτε να, τις, να έχετε και αντίτυπα. Το λέω αυτό γιατί αυτή η παρουσίαση είναι μακροσκελέστατη και απλώς κάποια σημαντικά σημεία θα ήθελα να παραθέσω εγώ που είναι και πολύ σχετικά με τη συζήτησή σας. Αν αναρωτιέστε ποιοι είμαστε, είμαστε μια εθνική μη κυβερνητική οργάνωση ε, χρηματοδοτούμε ε, από, αποκλειστικά από projects. Έχουμε δραστηριότητε σε διάφορου τομεί. Όταν ξεκινήσαμε, δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα, ε, δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με θέματα φύλου ή με διαφορά, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πολύ φλου έννοιε, πολύ αφηρημένε. Μετά από 6 χρόνια, καταλήξαμε να κάνουμε ακριβώ αυτά τα δύο. Να ασχολούμαστε δηλαδή με projects που έχουν να κάνουν με θέματα φύλου ή με θέματα διαφθοράς. Και σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε, όντως το θέμα της διαφορά στο Αφγανιστάν είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ό,τι αφορά τη διαφορά του Αφγανιστάν στην παγκόσμια κατάσταση. Στην ε, δικιά μας εργασία τα τελευταία 5 με 6 χρόνια έχουμε καταγράψει τέσσερις πυλώνες που εμποδίζουν την εξυγίανση του διαφορμένου συστήματος του Αφγανιστάν. Προφανώ η κυβέρνηση έχει να παίξει ρόλο. Προφανώ ο ιδιωτικό τομέα επίση επωφελείται σημαντικά από τη διαφθορά. Δεν είναι τόσο προφανέ το ότι υπάρχει ε, γενική ε, έτσι, ε, θέληση από τον λαό να πληρώνει αυτές τις, να δωροδοκεί μάλλον. Και τέλος, πάλι δεν είναι τόσο προφανές ε, δεν είναι τόσο προφανής ο ρόλος των δωρητών ε, στο Αφγανιστάν και ο τρόπος με τον οποίο δαπανούν τα χρήματά τους. Η Ευρώπη ε, περίπου ένα δισεκατομμύριο το χρόνο δαπανά για το Αφγανιστάν. Αυτός είναι ο λειτουργικός ε, επιχειρησιακός προϋπολογισμός. Τα 900 εκατομμύρια από αυτά βρίσκονται στο σκάνδαλο με την Καμπούλ Bank. Δεν λέμε βέβαια ότι η Ευρώπη δαπανά χρήματα με διαφερμένο τρόπο, αλλά ίσως αυτά τα χρήματα όντως φρενάρουν την εξυγίανση, τη μεταρρύθμιση ενός πραγματικά διαφθαρμένου συστήματος. Και θα κάνω και κάποιες προτάσεις ως προς αυτό. Μέλο, κομμάτι της έρευνάς μας, όταν ασχοληθήκαμε με το θέμα της διαφθοράς, ήταν ένα πολύ απλό εγχείρημα. Βγήκαμε στον δρόμο και ρωτούσαμε τους πολίτες με πόσους διαφορετικούς τρόπους σας έχουν ζητήσει να δωροδοκίσετε. Και μετρήσαμε 30. 30 εκφράσεις δηλαδή υπάρχουν ε, στην αφγανική γλώσσα για, το, για τον όρο δωροδοκία. Υπάρχει και ένας κατάλογος στις διαφανίες μου. Ε, μερικές είναι αρκετά διασκεδαστικές ως λέξεις. Ας πούμε, με το δικό μου πρόβλημα τι θα γίνει. Ή το αν χρησιμοποιήσω το στυλό μου για να γράψω, ε, πρέπει να με πληρώσεις. Έχω κάποια σημεία που θέλω να σας αναφέρω για αυτούς τους τέσσερις τομείς. Ε, ο, ιδίο είναι η, η ψυχή του λαού και οι διεθνείς δωρητές. Οι άλλοι δύο τομείς είναι η κυβέρνηση και ο ιδιωτικό ε, τομέα Θα τα αφήσω προς το παρόν και αν έχουμε χρόνο θα επανέλθω. Το κοινό είναι δεδεθειμένο να ικανοποιήσει ε, και να μην αμφισβητήσει την εξουσία πληρώνοντας αυτές τις, ε, αυτά τα ποσά. 30 χρόνια μαχών στο Αφγανιστάν με όλα τα επίπεδα δικαιοδοσίας να θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα ε, αυτό είναι προφανώς ένας πολύ φυσιολογικός μηχανισμός αυτοάμυνας. Δεν θα αλλάξει αυτό με εξαρτίες ευαισθητοποίησης, δεν θα αλλάξει αυτό με ομιλίες. Οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται να αντιμετωπίσουν την εξουσία. Υπάρχουν πολύ χαμηλές ε, ε, επιδιώξεις ή προσδοκίες από τους υπαλλήλους είναι εκεί, υπάρχουν στη θέση τους για να σε βασανίσουν, όχι για να σε βοηθήσουν. Αυτή είναι η γενική αντίληψη. Υπάρχει μια τάση να, υπο, να, να μειώνει κανείς ε, στο λιγότερο δυνατό της, ε, την σχέση που έχει με τους ε, ε, δημοσίους υπαλλήλους γιατί όποτε τους χρειάζεται δημιουργούνται προβλήματα. Επίσης το κάνει αυτό γιατί φοβούνται, φοβάται τη δίωξη, δεν θέλει να, να τον γνωρίζουν, θέλει να είναι αόρατος σε αυτούς που έχουν εξουσία και βρίσκονται σε επίσημες θέσεις. Αν πάει κανεί σε κάποιο οργανικό υπουργείο για να κάνει μια δουλειά, για να κάνει κάτι, αυτό που ο κλητήρα στην πόρτα σε στέλνει σε κάποιον άλλον, τον ενδιάμεσο. Ο ενδιάμεσο ξέρει πόσα πρέπει να πληρώσει κανένα τον κάθε υπάλληλο για να πάρει την άδεια που χρειάζεται, για παράδειγμα. Αν προσπαθήσει κανεί να το κάνει αυτό μόνο του, και εμεί το κάναμε, μπορεί να πάρει τρει εβδομάδε. Αν πάει μέσω του ενδιάμεσου, μπορεί να πάρει τρει μέρε. Αν πα μόνο σου, δεν ξέρεις και πόσο να πληρώσεις και σε ποιον. Ενώ αν πας στον ενδιάμεσο θα σου δώσει μια τιμή και θα πάρεις και την αδειά σου και θα γίνει και η δουλειά σου. Είναι πολύ θεσμοθετημένα λοιπόν όλα αυτά στο Αφγανιστάν. international... Πάμε τώρα στους διεθνείς ε, δωρητές. Τι μπορούν να κάνουν. Έχετε ακούσει όλο, όλοι τον όρο burn rate. Έχετε ακούσει όλοι τον όρο μηδενικό προπολογισμό. Ξέρετε ότι όταν τα χρήματα δίνονται από, διαφορε... από συγκεκριμένα κράτη-μέλη ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ω υπερεθνικό οργανισμό, τα χρήματα αυτά πρέπει να δαπανηθούν. Αλλιώ θα υπάρξουν συνέπειε. Αυτό έχει πραγματικά μεγάλε αρνητικές συνέπειε στην ε, αντιμετώπιση τη ε, διαφθοράς στο Αφγανιστάν. Γιατί τα χρήματα πληρώνονται σε οργανισμούς που δίνουν αναπτυξιακή βοήθεια και σχετικές υπηρεσίες, δηλαδή οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος ε, των εταιριών που έχουν να κάνουν με υπηρεσίες παροχής αναπτυξιακής βοήθειας. Πληρώνονται λοιπόν με βάση το κόστος τους. Αν δεν δαπανίσει κανείς τα χρήματα στο, το, το, το, του κόστους, δεν μπορεί να ε, ζητήσει έξτρα. Επομένως, δεν δίνει κανείς ε, δουλειά σε ανθρώπους που μπορούν να κάνουν ποιοτική δουλειά, δίνει κανείς, ε, ε, βάζει μάλλον σε αυτές τις θέσεις άτομα 24 χρονών κορίτσια για παράδειγμα που κάνουν τους, τις συμβούλους του, του 60χρονου υπουργού. Είναι μάταιο. Αλλά αυτά τα χρήματα δίνονται ανάλογα με τα άμεσα κόστη. Και ο υπεύθυνο επικεφαλής αυτή τη εταιρεία που κάνει τι υπηρεσίε αυτέ, που παρέχει τι υπηρεσίε αυτέ και μπορεί να, ε, να ε, χρεώσει παραπάνω και να διατηρήσει και το γραφείο του στις Βρυξέλλες. Είναι αυτό διαφθορά? Εγώ θα έλεγα ναι. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί να υποπτεύουν οι δολητέ τα λεφτά που δαπανούν, αλλά αν υπάρχει κάτι τόσο συστημικά λαθασμένο για το πώ κατα... κατα... κατανέμονται τα χρήματα, τότε κανένα, καμιά υποπτική δραστηριότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί ε, ουσιαστικά ε, αυτό αναιρείται. Επίσης, εγώ δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ την κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Όποια κατηγορία α, έχετε ακούσει για το Αφγανιστάν, κάποιο επιχείρημα έχει από πίσω. Αλλά μην ξεχνούμε ότι αυτό είναι και ο πιο εύκολο στόχο. Ο πιο δύσκολο στόχο είναι το πώ δαπανούμε τα χρήματα, τι βαθμό ελέγχου έχουμε για το πώ δαπανούμε τα χρήματα και επίση πρέπει να καταλάβουμε το φόβο του κοινού να προκαλέσει και να αμφισβητήσει την εξουσία και να αντιμετωπίσει την ε, διαφθορά. Το μόνο που ακούνε είναι ομιλίες από εμά, ενώ αυτοί είναι τελικά αυτοί που υποφέρουν από τη διαφθορά. Σε τι καταλήγουμε λοιπόν. Η αναδόμηση όχι μόνο στο Αφγανιστάν αλλά και σε, όλες, σε όσες χώρες έχουν θέματα με κατακαιρματισμένα συστήματα θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο έτσι ώστε κάποια στιγμή να ξεκινήσουν να έχουμε αποτελέσματα. Όχι με στρατηγικές ε, εξόδου το 2022 ούτε με αναμένοντας άμεσα αποτελέσματα σε 5-10 χρόνια. Για να προχωρήσουμε πρέπει να κατανοήσουμε το σύστημα. Για να κατανοήσουμε το σύστημα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Τα διάφορα μοντέλα που εισήχθησαν στο Αφγανιστάν, ε, έτσι όπως ας πούμε δούλευαν τα πράγματα στην Αφρική ή στην Κολομβία, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Κανένα από τα μοντέλα που, που εισήχθησαν στο Αφγανιστάν, κανένας δεν λειτουργήσε. Υπάρχουν ε, μονάδες ε, που ασχολούνται με θέματα φύλου σε κάθε Υπουργείο. Ε, έλυσαν τίποτα? Όχι. Είναι αυτός ο, τρόπος για να κάνουμε το gender mainstreaming? Όχι. Υπάρχουν εποπτικές αρχές που δημιουργούνται γιατί οι, όλες οι θέσεις γίνονται στην κυβέρνηση για την διαφθορά. Είναι πραγματικά ένα με το πρόβλημα αυτό και δεν λύνεται με ένα αναλυγητικό, Είναι πρόβλημα συστημικό να αλλάξουμε την πεποίθηση των ανθρώπων. Για να γίνει αυτό πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Για να αλλάξουν το σύστημα η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι λαμβάνει χρήματα από διάφορους διεθνείς οργανισμούς, η κυβέρνηση μπορεί να πει ότι δεν θέλω να αλλάξω εγώ τίποτα και το κάνει. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να σκεφτούμε άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά πέραν της κυβέρνησης. Βεβαίως να μην χάσουμε το τι γίνεται με την κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και άλλες διοικητικές δομές. Και πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα. Πρέπει να αλλάξουμε το μηδενικό προπολογισμό και την παγίδα αυτή που έχουμε βάλει. Πριν μιλούσαμε για την αναλλαγή της, ε, της νομοθεσίας από την κρατική σε την ομοσπονδιακή. Όλα αυτά είναι πολύ καλά, αλλά θέλουν και πόρους και χρόνο. Αυτό που σας λέμε είναι απλό. Πρέπει να κατανοήσουμε πόσα πληρώνουμε έναν ε, ε, ηλεκτρολόγο και έναν, ας πούμε υδραυλικό στην Καμπούλ. Ε, πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η τιμή του. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να του δίνουμε ό,τι λεφτά θέλουμε με ένα ανοιχτό πορτοφόλι, γιατί έτσι τον διαφύρουμε και αυτόν. Τι κάνουμε λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξή. Οι, διάφορες οργανισμοί, οι διάφοροι οργανισμοί που υπάρχουν τη ε, της ε, των πολιτών μπορούν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Μπορούμε να τους συμπεριλάβουμε ως προϋπόθεση για να αποδοθούν τα χρήματα στα ε, αφγανικά ε, υπουργεία πού βρίσκεται, πού θα συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών και πώς θα χρησιμοποιήσετε τα χρήματά μας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε. Επίσης, οι έρευνες που γίνεται. Πριν από λίγα χρόνια έκανα μια συζήτηση στις Βρυξέλλες με κάποιον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είπα ο προγραμματισμό σας πώς γίνεται και η έρευνα πώς γίνεται. Μου είπε δεν κάνουμε καμία έρευνα, απλώς κάνουμε προγραμματισμό. Και από πού μαθαίνετε, πού ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ξέρουμε, μου είπε. Ελπίζω να έχει αλλάξει αυτή η στάση. Και νομίζω ότι έχει αλλάξει μια που είμαι σήμερα εδώ. Τώρα, ε, δραστηριότητες μέσω των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων και άλλων ε, ανθρώπων από άλλες χώρες. Ε, και η Ελλάδα έχει διαφθορά. Ε, μάθει η, αυγανική η κοινωνία από την ελληνική πώ αντιμετωπίζεται η διαφθορά. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες, και Κένια και, και στην Ινδία ε, άνθρωποι που δωροδοκούνται ε, και ε, τους βιντεοσκοπούν και τους βάζουν στο διαδίκτυο. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν και για, την, για το Αφγανιστάν. Δεν κοστίζουν τίποτα υποστήριξη διαφόρων δραστηριοτήτων ε, για την, ε, μέσω ε, δραστηριοτήτων ε, επιτόπου, ας πούμε στην προσευχή της Παρασκευής, που είναι πολύ σημαντική. Ε, μια παρόμοια παρουσίαση είχα κάνει πριν από δύο χρόνια και κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν έχει την αντιμετώπιση της διαφοράς ως σημείο της, ε, της δουλειάς του ή της προεκλογικής του εκστρατείας. Δεν τους ενδιαφέρει, αλλά πρέπει να μάθουν να του ενδιαφέρει. Ε, επίσης, τα περιφερειακά φόρουμ και η Κεντρική Ασία έχει θέμα με την ε, ε, διαφθορά. Μπορεί να υπάρξουν λοιπόν συναντήσεις τέτοιες με ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και δεν κοστίζουν τίποτα. Μείωση της εξάρτησης από, τέτοιες, από εταιρείες που έχουν ε, παράνομα κέρδη. Επένδυση σε, στον προγραμματισμό με αποκεντρωμένο τρόπο, έτσι ώστε μια μεγάλη εταιρεία να μην παίρνει όλο το, όλο το, όλη τη χρηματοδότηση, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος και για τις τοπικές οργανώσεις να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί. Αυτά από μένα και ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Σίγουρα θα σημειωθούν δεόντως και από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Φιρντρόρη, που έχει και αυτός 15 λεπτά για να παρουσιάσει την ε, παρέμβασή του. Παρακαλώ αν μπορείτε να τηρήσετε το 15 λεπτό. Κύριε Ντόρη. Uh, Ευχαριστώ. Ε, ε, προέρχομαι από δύο οργανισμούς που αφορούν και τη διαφθορά και το περιβάλλον. Μία είναι η Λάγκα, ασχολείται με την καταπολέμηση της διαφθοράς και αντιδιαφθορά, δεύτερος οργανισμός που εστιάζεται επί της διαφθοράς εντός του τομέα της, ανα... των διαφόρων επιχειρήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Θα είναι κάπως ε, η διαδρομή μας άγρια ε, θα μιλήσω λοιπόν για το έγκλημα, θα μιλήσω για τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα που συνδέονται με την εγκληματικότητα στον τομέα της ε, Άγρες Πανίδας. Ας βγούμε από τις ψυχρές βρύξερες και ας πάμε στα δάση ε, τα τοπικά της Δυτικής Αφρικής. Βλέπετε υπέροχα πλάσματα εδώ, τους γορίλες βλέπετε, οι οποίοι τελικά θα εξαφανιστούν σε 15 με 20 χρόνια. Και αυτό λόγω ε, παράνομου εμπορίου πανίδας των ζώων. Και επίσης και των ελεφάντων που ζουν στα δάση. Η μοίρα δεν είναι διαφορετική. Ανακαλύψαμε την περασμένη εβδομάδα μέσω ε, έρευνας που έκανε αρμόδιος φορέας όπου χάσαμε πάνω από 60% των ελεφάντων των δασών την τελευταία δεκαετία και σε 10-15 χρόνια και αυτοί θα εξαφανιστούν και όλα αυτά λόγω του παρανόμου εμπορίου των ζώων, αγριών ζώων τα λιοντάρια. Ε, βασικά έχουμε 50% λιγότερα λιοντάρια από ό,τι νομίζαμε ότι είχαμε στον κόσμο. Στις περισσότερες χώρες που εργαζόμαστε τα λιοντάρια ήδη έχουν εξαφανιστεί ή πρόκειται να εξαφανιστούν στα επόμενα δύο χρόνια. Και όλα αυτά λόγω παράνομου εμπορίου αγρίων ζώων. Όσον αφορά το ρινόκερο, η ιστορία του δυτικού, που βρίσκεται στη Δυτική και Κεντρική Αφρική του Μαύρου Ρινόκερου, ήδη η μοίρα του έχει κρυθεί. Εξαφανίστηκε το 2007 λόγω παράνομου εμπορίου αγρίων ζώων. Η ίδια η φύση δέχεται επίθεση από το εμπόριο αυτό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό είναι το πρόσωπο του εμπορίου αυτού. Βλέπετε εδώ το πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου που πάει από Καμερούν προς Νιγηρία με τέσσερις μεγάλους ε, σάκους ε, ε, μαριχουάνας. Έχετε πάνω ένα δοχείο με κοκαίνη και στο μέσο, στο κέντρο της εικόνας, αν δείτε πολύ προσεκτικά, βλέπετε κάτι σε κάτι πάνες και αυτό είναι ένα, ένα, ένα μωρό πυθικάκι. Εδώ βλέπετε, συλλήφθη με το μωρό το πυθικάκι. Και αν αναρωτηθείτε τι κάνει τι κάνει το πιθηκάκι με τη μαριχουάνα και την κοκαίνη στο φορτίο αυτό. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι είναι σοβαρό θέμα το εμπόριο αυτό των ζώων. Είναι το πέμπτο σε τάξη παράνομο εμπόριο, είναι οργανωμένο έγκλημα, συνδέεται με το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Αν ακούσατε για την αύξηση του, της λαθροθυρίας των ελεφάντων, θα καταλάβετε ότι ε, έτσι εξηγείται και το ελεφαντοστούν, το εμπόριο το παράνομο ε, που έχει αυξηθεί μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια μπορούν να βγουν από το εμπόριο των χαβλιοδόντων. Λοιπόν, η μόνη δίωξη που έγινε όσον αφορά συνδικάτο παράνομου εμπορίου ε, ελεφαντοστού στο Καμερούν, στη συνεργασία με το Interpol. Βλέπετε εδώ κινητό σαρωτή, ε, εμπορευματοκιμώτιο 40 ποδών περίπου 10 μέτρων, 12 μέτρων. Έχετε, έχει δηλωθεί ξυλία που εξάγεται από το Καμερούν και πάει στο Χονγκ Κόνγκ, στο κέντρο. Αριστερά βλέπετε υπάρχει ένα ψεύτικο χώρος, κάτι πιο πυκνό φαίνεται σαν φορτίο, σκοτεινότερο. Θα δείτε ότι υπάρχει και κάτι αιχμηρό και είναι ελεφαντοστούν. 603 κομμάτια χαβλιοδόντων, 3,9 τόνοι. Και μια κατάσχεση ε, αυτού του προϊόντος σημαίνει ότι προέρχεται από 300 ελέφαντες που σκοτώθηκαν. Και αυτή τη δραστηριότητα την κάνουν κάθε δύο μήνες αυτή τη μεταφορά με τα ψεύτικα τμήματα, τα κρυμμένα τμήματα εντός του κοντέινερ. Από τη δεκαετία του 80 ε, το αυτή η οργάνωση. Ε, ανεπανόρθωτη ζημιά που έχει προξενήσει. Και μία μόνο παράνομη οργάνωση στη βιοπικιλότητα έχει προξενήσει τεράστια ε, ζημία. Συντόνιζαν πάρα πολλούς σε πολλές χώρες αυτοί. Πολλούς λαθροθύρες. Αυτή η κλιματική οργάνωση έπρεπε να ακολουθεί μια πολύ παρα πολλου σε πολλες χωρες αυτοι πολλου λαθροθυρες αυτη η ιεραρχία και προστασία που εφαρμοζόταν μέσω δικτύου διεφθαρμένων αξιωματούχων, στρατηγών, δικαστών, δημάρχων, υπουργών, μελών κοινοβουλίου. Αυτοί οι άνθρωποι επληρωνόταν από αυτή την παράνομη οργάνωση για να τους βοηθάει. Βέβαια, σχετίζονται και με άλλη παράνομη συνδυότητα ξέπλυμα χρήματο, προφανέστατο, σχέσει με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών μέσω Πακιστάν και υποθέτουμε και ότι συνδυόταν και με το εμπόριο όπλων διότι αυτά τα κυβότια ανακυκλωνόταν πήγαν από Αφρική, Ασία, από Ασία, Αφρική και λοιπά τα κοντέινερ και χρησιμοποιούνται για να φέρουν στην Αφρική όπλα, αλλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Και άλλα. Έγκλημα κατά της πανίδας. Εδώ έχουμε γκρίζους παπαγάλους, αθώα πουλιά, πολύτιμα για το παράνομο εμπόριο. Εδώ βλέπετε κλουβιά, περιέχουν αποστολή ε, παπαγάλων, περίπου χίλιους παπαγάλους που αξίζουν ένα με δύο εκατομμύρια δολάρια παράνομα κερδί. Στο Καμερούν αυτό γίνεται κάθε δύο εβδομάδες. Είναι πάρα πολύ κερδοφολα επιχείρηση. Και εντοπίσαμε ότι ο Γενικός Γραμματέας υπεύθυνο για την άγρια πανίδα στο Καμερούν, ο Υφυπουργός ουσιαστικά ήταν αναμειγμένος. Και άλλο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη αυτή εγκληματική οργάνωση γινόταν συνεχείς δωρές από αυτούς προς τα κόμματα της χώρας. Άρα υπήρχε κάποια πολιτική προστασία στον αφορά την παράνομη αυτή δραστηριότητα. Να σας δώσω τώρα κάποιες ελπίδες επίσης και με ποιους τρόπους μπορούν να καταπολεμηθούν τα προβλήματα αυτά και η διαφθορά σχετική. Η Λάγκα ε, είναι ο πρώτο, η πρώτη ΜΚΟ για την επιβολή του νόμου όσον αφορά την Πανίδα. Ξεκινήσαμε στη μηδέν, μηδέν διώξη στην Κεντρική και Δυτική Αφρική, άρα δεν εφαρμόστηκε ο νόμος καθόλου και είδαμε ότι το πρώτο εμπόδιο για να εφαρμοστεί ο νόμος είναι η διαφθορά. Σχετικά με την Πανίδα, έτσι η νομοθεσία. Προσπαθήσαμε να καινοτομήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο καταπολέμησης διαφθοράς και για να εφαρμοστεί ο νόμος. Όχι μόνο για την αγριαχλωρίδα και Πανίδα, αλλά γενικά να δραστηριοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών και να αλλάξει την πραγματικότητα όσον αφορά τη διαφθορά. Πώς λειτουργούμε τώρα. Συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεως και ΜΚΟ. Η ΜΚΟ διενεργεί έρευνες. Έχει αυτή την εντολή. Έχουμε διάφορους μυστικούς ε, ελεγκτές που δυσδύουν στα παράνομα δίκτυα, εντοπίζουν τους στόχους, τη διαφθορά, συμμετέχουμε σε διάφορες, διάφορες επιχειρήσεις συλλήψεων, παρακολουθούμε τις επιχειρήσεις, δίνουμε την νομική συνέχεια που δίδεται μέχρι την εκδίκαση της υποθέσεως, ε, παρακολουθούμε τη διαφθορά, την καταπολεμούμε, χρησιμοποιούμε τα ΜΜΕ για να δημοσιοποιήσουμε τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Είμαστε σωματοφύλακες ουσιαστικά της διαδικασίας επιβολής του νόμου. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι κάτι πραγματικό για μας. Στατιστικά στοιχεία σας παραθέτω. Μόνο το Καμερούν, αν δούμε σαν χώρα, πάνω από 500 επιτυχείς συλλήψεις έχουν επιτευχθεί, κυρίως πολλοί δημόσιοι αξιωματούχοι έχουν συλληφθεί. Από τα στατιστικά στοιχεία βλέπουμε ότι 85% της υποθέσεις έχουν, ε, εκεί έχουν τεκμηριωθεί προσπάθειες δωροδοκίας. Επίπεδο σύλληψης Άρα πώς να λειτουργήσει η αστυνομία όταν 85% των, 85 ε, των ε, περιπτώσεων δεν συλλαμβάνει και δωροδοκείται. Και δεν είμαστε εκεί να προσμετρήσουμε, αλλά να καταπολεμήσουμε. Καταπολεμούμε λοιπόν όλη αυτή την προσπάθεια διαφθοράς, κερδίζουμε για να συνεχιστούν οι ιδέες διαδικασίες. Το δικαστικό σύστημα δεν τα πάει καλύτερα. Στο 80% από τις 500 δικαστικές υποθέσεις που κερδίσαμε, στο 80% των υποθέσεων μπορώ να σας πω πώς θα ζητούσε ο δικαστής, πόση δωροδοκία ζητούσε. Σκεφτείτε πόσο δυσλειτουργικό, δυσλειτουργικό είναι το σύστημα όταν 80% των υποθέσεων ε, δεν καταλήγουν σε απόδοση δικαιοσύνης. Και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τις απόπειρες διαφθοράς ε, έξι χώρες από μηδέν διώξεις φτάσαν στο επίπεδο να φυλακίζεται ένας μεγάλος λαθρέμπορος ε, άγριας, αγρίων ζώων την εβδομάδα. Άρα αν ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω είμαστε πολύ αποτελεσματικοί. Πολλούς, πολλοί από τους φυλακισμένους είναι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι ψηλού επίπεδου και μπορέσαμε να εντοπίσουμε και να διώξουμε πολλούς ε, δικαστές. Και πάμε και σε άλλου τομεί. Εμπόριο παιδιών, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Πάμε και σε άλλου τομεί να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Και δείχνει αυτό πώ οι πρωτοβουλίε από κάτω προ τα πάνω, από την κοινωνία των πολιτών, μπορεί να είναι καινοτόμε πρωτοβουλίε και πιο αποτελεσματικέ. Όχι μόνο στην προσμέτρηση τη διαφθορά, αλλά στην καταπολέμησή τη και να κερδίζουμε μία υπόθεση κάθε φορά. Όλα αυτά είναι καλά και ωραία γιατί, τι τη νοιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, γιατί ό,τι συμβαίνει στο, άγριο, στο, στη ζωή στην Αφρική συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, και φτάνουν, ας πούμε, βλέπουμε του παπαγάλου που έρχονται από την, ε, στην Ανατολική Ευρώπη και πάνε στη Δυτική. Έχουν αναμειχθεί η Ολλανδία και η Τσεχική Δημοκρατία και ε, ε, το παράνομο μπορεί όσον αφορά τους πίθηκους και τους μεγαλοπίθηκους φτάνουν μέσω αέρα και θάλασσας. Το είδαμε και εδώ. Όπου συλλάβαμε έναν ε, που είχε παραδεχτεί ότι είχε πουλήσει πάνω από 500 πυθίκους. Κάναμε προβολή και είδαμε ότι τελικά πρέπει να σκοτωθήκαν πάνω από 5.000. Αυτό το άτομο το συγκεκριμένο εξήγησε το πώς πολλούνται πούλησε και εξήγαγε πέντε πίθηκους πάνω σε πλοίο. Στείλαμε αυτές τις πληροφορίες στις Ισπανικές Αρχές και μέσω του Ίντερπολ. Και κλιπαρίσαμε να κάνουν κάτι. Είπαμε έχετε δύο μήνες να προετοιμαστείτε για να συλλάβετε τον ένοχο που θα φτάσει στις ακτές σας. Δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα από την Ισπανία. Άλλο θέμα για το εμπόριο ελεφαντοστού. Παρόλο που το ελεφαντοστούν φτάνει στην Κίνα και στην Ασία, το μεγαλύτερο ποσοστό και κάποια από αυτά, κάποια από αυτά φτάνουν στην Ευρώπη. Σύλληψη ενός μεγάλου εμπόρου στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έλαβε χώρα, όπου αυτός έδωσε πληροφορίες για το πώς αυτοί τακτικά εμπορευόταν και έστελνε ελεφαντοστούν στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Μας έδωνε συγκεκριμένους τόπους όπου βρισκόταν αποθέματα και στην Ιταλία και στη Γαλλία Λοιπόν, δείξαμε συνεργασία, στείλαμε τις πληροφορίες μέσω Interpol Επίσης, η μόνη απάντηση που είχαμε ήταν ότι οι δυνάμεις που είναι υπεύθυνε για αυτά τα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν επαρχική στελέχωση και δεν έχουν και εντολή και το ένταλμα έρευνας για να βρουν αυτό το εμπόρευμα. Και δέρματα τομάρια λονταριών από το Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και Κονγκό και πού πάνε αυτά τα δέρματα. Μέσω Γαλλίας και Βελγίου πηγαίνουν, περνούν αυτά τα δέρματα μέσω κυνηγών σαφάρι που συμμετέχουν στη σαφάρι. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, έχει αποτρεπτικά ε, μέτρα για να εμποδίσει το εμπόριο. Είναι παράδεισος για αυτά τα εμπορεύματα. Σε κάθε χώρα που εργαζόμαστε συλλαμβάνουμε έναν ένοχο μια φορά την εβδομάδα. Αν πάρουμε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα ότι ο αριθμός των εγκληματιών που μπαίνουν στη φυλακή ε, μετρώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Πολύ ήπιες οι ποινές, δεν προβλέπεται φυλάκιση, σχεδόν ποτέ. Ε, ελάχιστος μεθοριακός έλεγχος εφαρμόζεται και υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες ξεπλήματος χρήματος. Βασικά το μήνυμά μου ποιο είναι. Έχω εδώ το σχέδιο έκθεση στα χέρια μου. Ε, όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς και του ξεπλήματος χρήματος. Καμία λέξη εδώ για το έγκλημα στον τομέα του εμπορίου του παρανόμου των αγρίων ζώων, που είναι πέμπτο σε επίπεδο παράνομου εμπόριο στον κόσμο και έχει φοβερές συνέπειες όσον αφορά φοβερά αποτελέσματα. Εμπλέκονται κάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι παράδεισος για αυτό το εμπόριο και πρέπει αυτό αυτός ο τομέας αναφέρεται στην έκθεση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν ποινές που θα έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Συμβαίνουν όλα αυτά στην Αφρική και θα συμβούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σωστά αποτελέσματα. Μπορούμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα ελέγχου που τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναφέρουν τι γίνεται με τις διώξεις. Αυτό συμβαίνει στην Αφρική. Αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο για το έγκλημα κατά των αγρίων ζώων, μπορούν να γίνουν όλα αυτά για όλα τα είδη διαφθοράς. Να ασκήσουμε θετικές πιέσεις με αυτόν τον τρόπο επί των κρατών μελών. Ε, και βέβαια χρειάζεται αύξηση του αριθμού. Χρειάζεται καλύτερη στελέχωση αστυνομία. Θα ήθελα να αναφέρω και κάτι άλλο για τι ευθύνε που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διασύνδεση όσον αφορά με ε, το θέμα τη αναπτυξιακή βοήθειας. Παράλληλα με το έγκλημα κατά των αγρίων ζώων και του περιβάλλοντος, βλέπουμε τι γίνεται στο Καμερούν, αντίδραση υπήρξε σφαγή ελεφάντων στο Καμερούν έλαβε χώρα. Υπήρξε αντίδραση και οδήγησε σε αύξηση της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. βρέχει χρήματα λόγω της καταστροφής, λόγω ελλειπούς ε, πλημελούς διακυβέρνησης. 2,5 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν γρήγορα για προγράμματα σε μικρή περιοχή, 1,5 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν για συνεδριάσεις, όχι, την κυβέρνηση και 1,8 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν για συνεδριάσεις εντός 45 ημερών έπρεπε να δαπανηθούν. Αποτέλεσμα όλων αυτών, αποτέλεσμα της ταχείας χρηματοδοτήσεως, ένεσης χρημάτων, λειτουργεί σαν καύσιμο που ρίχνεται στη φωτιά σε ένα διεφθαρμένο σύστημα. Θέλαμε να, να επιληθεί ένα πρόβλημα δυναμικού, ενώ το πρόβλημα ήταν διακυβέρνησης. Αντιπαραγωγική την η χρηματοδότηση μπορούν να ληφθούν πιο έξυπνες αποφάσεις για τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να ελαχιστοποιείται η διαφθορά, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και η κοινωνία των πολιτών μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο λόγο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κύριε Τρόντι, Πραγματικά μας προβληματίζουν αυτά που είπατε. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω, ε, βλέπω ότι δεν έχετε βάλει τα ακουστικά σας, δεν έχετε βρει το κανάλι, οπότε θα τα πω και στα αγγλικά. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι μας εκπλήσει κατά κάποιο τρόπο. Ίσως γιατί είμαστε αφελείς, παραμένουμε αφελείς, πάντως μας εκπλήσει και μας σοκάρει. Πολύ μεγάλο μέρος αυτών που είπατε. Στην Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα χαρούμε πάρα πολύ να μας στείλετε συγκεκριμένα στοιχεία για αυτά τα οποία καταγγέλλετε και να είστε βέβαιος ότι θα αναλάβουμε δράση για τα, τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην τελευταία ομιλήτρια αυτής της Τρογγυλής Τράπεζα, την κυρία Πέτρα Κνόιερ, που όπως προείπα είναι διευθύντρια της Όλαφ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας και τα πολέμης απάτης. Πάρα πολύ ε, γνωστού και σεβαστού φορέα ε, στο κοινοτικό πλαίσιο διότι χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο θάρρος και τόλμη. Πολύ συχνά γύρει ζητήματα που μπορεί να αφορούν και άκρος ισχυρούς ε, ανθρώπους ή φορείς και πρέπει να παροτρύνουμε την ε, Διευθύντρια να συνεχίσει ε, προς την κατεύθυνση. Θα σας ακούσουμε κυρία Κνόρη με τη μάγιστη προσοχή. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Good morning, Mr. Lee. Good morning, Mr. Καλημέρα σας, κύριε Μαρτίνες, κύριε Νιτοντάν, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω ε, τις ευχαριστίες μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως προς την κυρία Εύα Ζολή για την πρόσκληση που μου δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον φόρουμ ε, στο οποίο τίθεται το ζήτημα της διαφθοράς σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος ε, και το οργανωμένο έγκλημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλώ εξ ονόματος της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της ΑΠΑΤΗ την οποία είμαι διευθύντρια από το Δεκέμβριο του 2012 και είμαι αρμόδια για τις έρευνες σε σχέση ακριβώς με τον τομέα αυτό. Όπως γνωρίζετε, η Όλαφ είναι ένας πολύ σημαντικός ε, πρωταγωνιστής ε, λόγω των ερευνών που αναλαμβάνει για την ε, καταπολέμηση της διαφθοράς. Και στόχος είναι τα επιχειρησιακά μας αποτελέσματα να είναι όλο και πιο αποτελεσματικά. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να αναφέρω ότι είμαι και εισαγγελέα και διατέλεσα τα τελευταία πέντε χρόνια μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη. Το Ζαν Πιέρ Μπεγκόμπο, παραδείγματος χάρη, τον τέος αντιπρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, διέπραξε ιδεχθή εγκλήματα, ε, τον ε, δίκασε και ήμουν και εισαγγελέας στη Γερμανία κατά το παρελθόν. Ήμουν και εισαγγελέας. Μου ζητήθηκε να σας παρουσιάσω τις εμπειρίες της Όλαφ για την πρόληψη αλλά και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχει σημασία η διαφθορά, γιατί πρέπει να την καταπολεμήσουμε, να την αποτρέψουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η διαφθορά εκτιμάται ότι θα κοστίσει στους Ευρωπαίους φορολογούμενους 120 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το 1% δηλαδή του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παρούσα η διαφθορά σε όλες σχεδόν τις χώρες και έχει άκρως καταστροφικά αποτελέσματα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, διότι παρεμποδίζει οποιαδήποτε ανάπτυξη, οικονομική μεγέθυνση και δημοκρατία. Τέσσερις, στους πέντε Ευρωπαίοι πολίτες υποστηρίζουν ότι η διαφθορά είναι μείζον πρόβλημα στις χώρες τους και υπογραμμίζουν έτσι την ανάγκη μιας πιο στεναρής πολιτικής δέσμευσης για την αντιμετώπιση του κλίματος αυτού που προκαλεί οικονομικό-κοινωνικό κόστος. Οι δωροδοκίες, ε, οι παράνομες ε, πληρωμές ε, παρακάμπτουν τις δημοκρατικές διαδικασίες, παρεμποδίζουν την εύθυμη λειτουργία της οικονομίας και ουσιαστικά ε, είναι σε βάρος των ε, τίμιων συμπολιτών μας. Δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς μονοπόλιο των ε, βιομηχανικών χωρών, ούτε οι συνταγές που ισχύουν σε ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν κατά ανάγκη να εφαρμοστούν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όλο και περισσότερο οι αναπτυσσόμενες χώρες εκφράζουν το, την αποφασιστικότητά τους να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, απηχώντας διεθνείς πρωτοβουλίες όπως είναι η πράξη του Συμβουλίου του Μαΐου του 1997. Στις περισσότερες αψώνες χώρες υπάρχει άκρος διαδεδομένη διαφθορά. Είναι καθημερινότητα. Η κοινωνία έχει μάθει να ζει με τη διαφθορά. Ίσως δε μπορεί και να τη θεωρεί ένα στο τμήμα της κουλτούρας της χώρας. Υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί που βοηθούν στη διάδοση της διαφθοράς και την καθιστούν ε, συνήθη πρακτική στις αναπτυσσόμενες αυτές χώρες. Ουσιαστικά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημόσια λειτουργία αλλά και ιδιωτικοί φορεί λειτουργούν. Αυτό το πλαίσιο δημιουργεί τη διαφθορά. Η δημόσια διοίκηση στι αναπτυσσόμενε χώρε είναι συχνά γραφειοκρατική και αναποτελεσματική ενώ δε υπάρχουν πολλοί και πολύπλοκοι κανονισμοί ε, συνοδευόμενοι με, από ανεπαρκείς ελέγχους. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των αναπτυσσόμενων χωρών και ε, αυτά τα εκμεταλλεύονται, ε, τα εκμεταλλεύονται κυκλώματα διαφθοράς. Άρα υπάρχουν άλλα στοιχεία που οδηγούν στην διαφθορά σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει ένα σημαντικός παίκτη στο διεθνή στίβο για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Και είμαστε πρωτοπόροι γιατί έχουμε δημιουργήσει υπερεθνικά νομικά μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερο εταίρο, μάλλον δωρητή σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίω ό,τι αφορά τη βοήθεια που παρέχουμε σε αναπτυσσόμενε χώρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών τη, είναι ο ηγετικό δωρητή. Πάνω από το 50% του συνόλου των 53 δις ε, αναπτυξικής βοήθειας είναι το τελευταίο στοιχείο που έχουμε στη διάθεσή μας για το 2012, χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος ε, ε, από τη διαφθορά. Οι θεσμικές πολιτικές αδυναμίες των χωρών στις οποίες επενδύονται μεγάλα ποσά δεν θα πρέπει να υποτιμώνται. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σωστό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου τον τρόπο με τον οποίο θα πάνε οι πόροι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια βασική ανάγκη πλέον. Κυρίε και κύριοι, όπως όλοι γνωρίζετε, η Όλαφ έχει το καθήκον να καταπολεμά τη διαφθορά και την απάτη. Και αυτό περιλαμβάνει ταυτόχρονα και την πρόσπιση των συμφερόντων του, του προπολογισμού της Ένωσης. Χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να βεβαιώσουμε τις παρατυπίες που έχουν ε, να κάνουν με την ε, χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Διεξάγουμε έρευνες ε, βέβαια και σε τρίτες χώρες χρησιμοποιώντας τα νομικά μέσα που τρέπουν στην Όλαφ να έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες ώστε να βεβαιώσει τις παρατυπίες αυτές. τι συνιστά απάτη και ποια είναι η σχέση απάτης διαφθοράς. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα παρατυπιών που εντόπισε η Όλαφ και που οι αξιόλογοι συνάδελφοί μου προανέφεραν. Δίπλη χρηματοδότηση, τιμολόγηση, ε, φουσκωμένα τιμολόγια, δωροδοκίες, ε, πολλαπλή διόχη κτλ. Η διαφθορά, η διαφθορή είναι σημαντική για να συγκαλύψει ε, την απάτη και η απάτη είναι σημαντική για την ανάκτηση του κόστου της διαφθοράς. Με άλλα λόγια, η διαφθορά είναι ένα ακόμη μέσο που μπορεί να συγκαλύψει την απάτη για, να, για την απόκτηση παρανόμως ενός κομματιού του κοινοτικού προϋπολογισμού που έχει δοθεί ως χρηματοδότηση. Να σας δώσω κάποια εύγλωτα παραδείγματα. Μια Ευρωπαϊκή ΜΚΟ ε, για αποναρκοθέτηση σε μια χώρα που ήταν ε, ε, αντικείμενο πολέμου, φιλικού πολέμου, πήρε κάποια ποσά έπρεπε να έχει το απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και το προσωπικό. Και επίση έπρεπε να χαρτογραφηθούν οι περιοχές αυτές. Τι έδειξε η έρευνα τη Όλαφ. Η δικαιούχος ΜΚΟ για να μειώσει τις δαπάνες είπε ότι ανείχνευσε μεγαλύτερες περιοχές από αυτές που αποναρκοθέτησε τελικά. Άρα έβαλε σε κίνδυνο τις ζωές ανθρώπων. Οπότε μπαίνει σε δεύτερη μοίρα εδώ το οικονομικό, οικονομική χασούρα. Οι επιβλέποντες λοιπόν δεν έκαναν το σωστό έλεγχο. Η συγκάλυψη αυτών των ε, δραστηριοτήτων κατέστη δυνατότητα να αρχίσαμε εμείς να ερευνούμε την υπόθεση. Είδαμε ποιε είναι οι οικονομικέ ζημίες για τον προπολογισμό και υπήρξε και κοινοποίηση προ την ΜΚΟ στο πλαίσιο του συστήματο έγκυρη περιοδοποίηση και συναγερμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά άλλε πτυχές, η Όλαφ με την έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει περαιτέρω πορίσματα. Γιατί, γιατί οι συνθήκε στη χώρα δεν το επέτρεπαν. Δεν μπορέσαμε δηλαδή να βρούμε ποια ήταν η τελική αλήθεια κάποιες φορές δεν έχουμε την απαιτούμενη συνεργασία από τις ε, χώρες. Αν δείτε ένα τέτοιο σήμα, μια τέτοια πινακίδα, ε, κρύβεστε, τρέχετε, τρέχετε να κρυφτείτε, αν δεν το δείτε είστε ασφαλείς. Δυστυχώς χάρη στη διαφθορά δεν ήταν ασφαλής η ζωή πολλών πολιτών, γιατί δεν τοποθετήθηκαν αυτές οι πινακίδες εφόσον δεν ελέγχθηκαν όλες τις περιοχές που έπρεπε. Σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Η βοήθεια εδώ χορηγήθηκε μέσω ενό διεθνού οργανισμού που στη συνέχεια παρήχε άμεση δημοσιονομική στήριξη σε μια τρίτη χώρα που τελικά χρησιμοποιούσε ΜΚΟ, τοπικές και διεθνεί εταιρείε για την ανέγερση κάποιων εγκαταστάσεων για την παροχή εξοπλισμού και φαρμάκων. Ουσιαστικά στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα άσπτο εργαστήριο. that we the... Αποστηρωμένο εργαστήριο. Εδώ βλέπετε τις αρχές εργασίες ανέγερσης του εργαστηρίου. Δείτε απλά τις εικόνες και φτιάξτε εσείς ε, στο μυαλό σας την εικόνα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αφού καταβλήθηκα τα χρήματα. Τρία χρόνια συγκεκριμένα μετά. Αποφασίστε εσείς αν αυτό θεωρείτε ότι είναι ένα άκρος αποστηρωμένο ιατρικό εργαστήριο που θέλετε να επενδύσετε τα χρήματά σας αυτό ή που μπορεί να στείλετε τα παιδιά σας ή μέλη της οικογένειάς σας εκεί για θεραπεία. Φαντάζομαι ότι πολύ, δέκα φορές ε, πιο υγιεινό είναι το πάτωμα στα σπίτια σας από αυτό που βλέπετε στην εικόνα. Θα ήθελα τώρα να στρέψω την προσοχή σας ε, στο δεξί κάτω μέρος της εικόνας. Δεν ξέρω αν αναγνωρίζετε αυτό. Εκεί είναι μια πόρτα. Στη χώρα αυτή η θερμοκρασία είναι γύρω 40 βαθμούς. Φαντάζεστε ότι τα φάρμακα ε, θα έπρεπε να αποθηκεύονται σε μέγιστη θερμοκρασία 6 βαθμών. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται λόγια εδώ. Για δείτε το πίσω μέρος ε, στο κτίριο. Βλέπετε κάποιο είδους air condition, κλιματισμού που υποτίθεται ότι φροντίζει την αποθήκευση, να είναι σωστή σε συνθήκες αποθήκευσης των φαρμάκων. Εδώ βλέπετε ότι όταν πλέον ε, διατίθεται προς απόρριψη τα, τα φάρμακα, τα έτρωγαν ε, ποντίκια, μπαίνανε και στα υπόγεια ύδατα. Φυσικά για να έχουμε τέτοια κλίμακα διαφθορά πρέπει να υπάρχει και συνεργασία από τις αρχές. Πολλές φορές βέβαια δεν υπάρχουν ε, δυνατότητες και μέσα για την ε, έρευνα. Η Εθνή Οργάνωση τώρα που ήταν ο πρώτος αποδέκτης της δικής μας χρηματοδότησης στην προκειμένη περίπτωση ακολούθησε μια καινοφανή προσέγγιση. Δηλαδή δημοσιεύει τα πορίσματα, εταιρείε, ονόματα δημοσίων αξιωματούχων στο διαδίκτυο. Ο στόχος άσκηση πίεσης και μείωση της διαφθοράς για άλλα project. Εμείς όμως δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση γιατί πρέπει να τηρούμε τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πώς θα βελτιώσουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι την αποτελεσματικότητα που ε, μπορούμε να έχουμε στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε τρίτες χώρες. Θα ήθελα να σας διατυπώσω ορισμένες προτάσεις. Πρώτον, καλύτερη ροή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών, φορέων που δραστηριοποιούνται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους ε, οικονομικούς δωρητές. Υπάρχει ένα εργαλείο πληροφορικής, το Transparent Aid, όπως λέγεται, είναι σε εξέλιξη ανάπτυξη του αυτή τη στιγμή. Ε, αυτό θα βοηθήσει να έχουμε αποφυγή διπλής χρηματοδότησης του ίδιου project, για παράδειγμα. Τρίτον, είναι σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση Στι πληροφορίε, στην ενημέρωση. Μόνο έτσι όλα μπορεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Και αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη πολιτικών. Για παράδειγμα, ε, για τους πληροφοριοδότες. Τέταρτον, πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή θεσμική θέση. Γιατί σε έναν βαθμό η συνεργασία θα εξαρτηθεί από την πραγματική συνεργασία που υπάρχει όταν ανακύψει υπόθεση διαφθοράς ή απάτης. Αν υπάρχει λοιπόν μείζον δέσμευση μεταξύ όλων των εταίρων, και Επιτροπή, Κοινοβούλιο, ΑΕΔ, όλοι αυτοί πρέπει να στηρίξουν την Όλαφ. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τις πολύ δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται ορισμένες έρευνες της Όλαφ είναι να μην μιλήσω και για προσωπικό κίνδυνο που διατρέχει το προσωπικό τη όλα σε ορισμένε περιπτώσει. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου δηλώνοντα ότι η καταπολέμηση τη διαφθορά έχει γίνει πλέον μια πραγματικά παγκόσμια προσπάθεια. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι από το πόστο μας ο καθένας για να ποινικοποιήσουμε την προσφορά, την επαγγελία ή την α, παρότρινση και να διευκολύνουμε τη δίμευση, κατάσχεση και ανάκτηση των προσόδων από διαστηριότητες διαφθοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κνόιερ. Να είστε βέβαιοι ότι τουλάχιστον από πλευρά Ευρωκοινοβουλίου και από πλευρά Επιτροπής ανάπτυξη. η Όλαφ μπορεί να έχει την απόλυτη στήριξή μας. Γιατί εκτιμούμε και την αποτελεσματικότητά σας αλλά και την αναγκαιότητα, την ανάγκη της ύπαρξής σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους βουλευτές Δυστυχώ δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα, γι' αυτό θα σα παρακαλέσω στι παρεμβάσει να είστε όσο το δυνατόν πιο περιεκτικοί. Ο πρώτο που ζήτησε το λόγο είναι ο κύριο Νιτοντάμ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Ο κύριος που μίλησε για τα άγρια ζώα, πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Αν σα δίναμε ένα μαγικό ραβδί Ποιο μοναδικό πράγμα θα θέλατε να κάνει αμέσω η Ευρώπη, ή δύο-τρία αν θέλετε. Αλλά αν θέλατε να γίνει κάτι αμέσω, προτείνατε κάποια πράγματα. Ευχολόγιο θέλουμε, θα μα βοηθούσε. Για την κυρία τη Όλαφ. Το τελευταίο που ανέφερε με παραξένεψε. Πρέπει να ποινικοποιήσουμε τη δωροδόκηση. Καλή ιδέα. Αλλά δεν υπάρχει ποινική, ποινικό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώση, αλλά επίπεδο κρατών μελών. Άρα συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να υπάρξει ένα ποινικό καθεστώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αστυνομικό σώμα, δικαστήρια, φυλακέ κλπ. Χρειαζόμαστε ομοσπονδιακό επίπεδο αντιμετώπιση του εγκλήματο. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Α κάνουμε ένα γύρο παρεμβάσεων και ο καθένα από εσά μπορεί να απαντήσει. Δεύτερον, έχει το λόγο η κυρία Ματεουγιούμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρία Πρόεδρε. Οι τρεις παρεμβάσεις ήταν πυκνότατες, εμπεριστατωμένες, άκρως ενδιαφέρουσες. Στην πρώτη δεν την πρόλαβα. Ψήφισα στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Και με λυπεί το ότι δεν ε, ήμουν παρούσα στο πρώτο κομμάτι της ακρόασης. Ο κ. Πάρτο μίλησε για το Αφγανιστάν είναι αποτυχία των όσων προσπαθούσαμε να κάνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγα το 2008 στο Αφγανιστάν σε μια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού και είδαμε επιτόπου τι προσπαθούσε να κάνει η Ένωση. Είχαμε κονδύλια για να επιβληθεί τελικά κοινοβουλευτική δημοκρατία, να γίνει κάτι για το κοινοβούλιο. Θέλαμε να ε, βελτιωθεί αμοιβή των δικαστών και της αστυνομίας για να περιορίσουμε τη διαφθορά. Μας λέτε όμως τελικά ότι η διαφθορά έχει θεσμοθετηθεί πλέον, έχει γίνει θεσμός. Τα εργαλεία που είχαμε εφαρμόσει τότε εξυπηρέτησαν ή όχι. Τα εργαλεία λοιπόν που δημιούργησε η Ένωση τι έκαναν οι δωρήτριε χώρε, κυρίω η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, είχαν υποχρεώσει τον Καζάι να βάλει παντού ελεγκτές, ούτως ώστε οι δομές σε επίπεδο χώρας, περιφερειών, ότι λογοδοτούσαν. Δεν ξέρω αυτοί οι ελεγκτές υπάρχουν, εργάζονται και οι αναφορές που δίνουν είναι, δείχνουν την πραγματικότητα, επικρατεί διαφάνεια, έχω την εντύπωση ότι όχι και για το θέσω απευθυνόμενο προς την Εύα. Ε, υπάρχει χαλιναγώγηση τουλάχιστον των ελέγχων κλπ. Αποτυχία λοιπόν η συνεργασία με την κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Πλήρης αποτυχία. Εμείς σαν Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι ακόμα. Αλλά είναι πολύ απογοητευτικό. Κύριε Ντορή, δίκιο έχετε αυτό που συμβαίνει όσον αφορά την πανίδα που εξαφανίζεται. Είναι πραγματικά λυπηρό. Η σύμβαση ΣΥΤΕΣ έλαβε κάποια μέτρα που δεν αρκούν. Και οι χώρες προς Ανατολάς ενδιαφέρονται, έχουν συμφέροντα όσον αφορά το Elephant κατέστρεψαν αυτή την πανίδα που αποτελεί κομμάτι της βιοπικιλότητας. Κρίμα. Ακούσαμε την έκκλησή σας. Δεν θα μιλήσω ονόματι του συγγητού. Ίσως όμως κάποιοι από εμάς μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες. Εξαφανίζεται μια κληρονομιά. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει πολλή λαθροθυρία για είδη που δεν εξαφανίζονται, αλλά όσον αφορά τα μεγάλα ελαφοειδή. Και οι δασοκόμοι καταστρέφουν αυτά τα είδη. Η κυρία Μπαρντό έκανε μάχη στο πλευρό των κυνηγών που θέλουν να διατηρηθούν αυτά τα είδη των ελαφιών. Τα ελαφοειδή λοιπόν σε κάποιες περιοχές εξαφανίζονται λόγω των δασοκόμων που βλέπουν το δάσος σαν κάτι που έχει πιο πολύ οικονομική χρειά και όχι σαν ένα κομμάτι της βιοπικιλότητας. Ή θα σας πω κυρία ότι οι φωτογραφίες που μας δείξατε είναι φρικτές και οι λύσεις που μας προτείνατε είναι καλές. Αυτό που δεν κατανοώ είναι πως στην περίπτωση του εργαστηρίου που μας δείξατε ότι δεν οικοδομείται σε μία μέρα το εργαστήριο. Πώς δεν διαπιστώθηκε αυτό πιο νωρίς. Θα χρειάστηκε ίσως ένας χρόνος, δύο χρόνια για να κατασκευαστεί το εργαστήριο. Γιατί εκ των υστέρων υπήρξε αντίδραση. Αλήθεια, κανεί δεν αρνείται ότι η διαφθορά και σε αυτές τις χώρες περισσότερο από ό,τι σε εμά, είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς, γιατί δεν πήγαμε εκεί να κάνουμε μια επαλήθευση. Να δούμε ότι η κατασκευή ανταποκρινόταν στις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει. Μήπως έχουμε και εμείς κάποιες ενοχές, μήπως αμαρτήσαμε σε κάποιο βαθμό και εμείς. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριος Τάις Μπέρμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις σας. Ήταν πραγματικά συνεργαστικές, πολύ ενδιαφέρουσες. Ένα ερώτημα για τον κύριο Πάρτο. Είπατε ότι η διαφθορά υποκινείται και από την ανάπτυξη και ότι αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα στο Αφγανιστάν. Έχουν φύγει πολλά, πολλές δεκάδες εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων μάλλον στο Αφγανιστάν και αυτό οδήγησε σε τεράστια διαφθορά που δεν υπήρχε πριν από το 2001. Μετά το 2014 εσείς τι περιμένετε να γίνει, όταν θα είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα που θα εισραίουν στη χώρα, όταν θα έχουν φύγει οι στρατιωτικές δυνάμεις, ένα μεγάλο μέρος αυτών, αυτό δεν θα έχει ε, συνέπειες στο μέλλον της χώρας. Εσείς τι περιμένετε. Ποια πολιτική περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε αυτό το νέο τοπίο μετά το 2014 σε σχέση με τη διαφθορά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Τάις. Ο κύριος Γιακολίνο που είναι και εισηγητής για το θέμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε το σχόλιο του. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε τρεις παρεμβάσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Αναφέρθηκαν κάποιοι ρόλοι πολύ σημαντικοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει πόρους 53 δισεκατομμύρια ευρώ αναφέρθηκε στις αναπτυσσόμενες χώρες το 2011. Πολύ μεγάλο ποσό. παίζουν ρόλο οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και τρίτε χώρε. Καθένα από του φορεί έχει ευθύνε και ρόλο. Είναι σημαντικός ο ρόλος της μεγάλης ε, γραφειοκρατίας της αδύναμης δημοκρατίας. Η κυρία Γνέρ είπε ότι είναι πολύ σημαντική ανταλλαγή πληροφοριών για τη συνεργασία. Ερώτηση και σκέψη για τους τρεις προσκεκλημένους. Ίσως θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες αυτές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Να, ε, να εξετάζονται καλύτερα πριν τους διατίθενται πόροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να γίνει επιμερισμός των ευθυνών Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των χωρών. Και χρειάζονται και ισχυρές μεγάλες κυρώσεις. Ερώτηση λοιπόν για την κυρία της Όλαφ. Τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με αυτά τα χρήματα που διατίθενται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα, ορίστε. Eh, Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μου λένε ακόμα, δεν μου έχουν πει ακόμα το όνομα, τέλο πάντων θα μου πούν ε, σε ποιον εκπρόσωπο δώσω το λόγο, αλλά ήθελα και εγώ να επιμείνω για να δω και την αντίδραση των συναδέλφων. Ε, θα ήθελα να επιμείνω σε κάτι που είπε έτσι εν παρόδο, είχα πει στην αρχή, δηλαδή ότι σε ποιο βαθμό η διαφθορά είναι επικίνδυνη για την αναπτυξιακή συνεργασία. Γιατί πρέπει να έχετε όλοι σας υπόψη, όπως εμείς το έχουμε υπόψη μας, ότι σε, ένα, σε μια χρονική περίοδο που υφίστανται σημαντικούς, σημαντικές περικοπές ή προπολογισμοί, η αποτελεσματικότητα των δράσεών μας είναι και το επιχείρημα για την, ε, τις λιγότερες ή τις περισσότερες περικοπές. Δηλαδή, αν είναι αναποτελεσματική η δουλειά μας, όπως φαίνεται να προκύπτει από ορισμένε παρεμβάσεις, αυτό δίνει επιχειρήματα μεταξύ άλλων στα κράτη-μέλη για να προτείνουν περικοπές, πολύ σημαντικές περικοπές σε αυτό τον τομέα που είναι ε, λίγο πιο μακρινός, άρα έχει μικρότερη ευαισθησία σε σχέση με άλλα κεφάλαια του προπολογισμού που άπτονται άμεσα τη καθημερινότητα των πολιτών. Άρα είναι θέμα αποτελεσματικότητα και του ε, πόσο η διαφθορά επηρεάζει. Αν επηρεάζει λίγο, ε, έτσι θα μπορέσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη της κυβέρνησης, αλλά και τους πολίτες. Αυτές οι φωτογραφίες που μας έδειξε όλα, για παράδειγμα, και αυτά τα στοιχεία θα κάνουν τους πολίτες που χρηματοδοτούν τέτοιου είδους δράστα να σκεφτούν ότι άλλοι μηχανισμοί χρειάζονται. για να μπορούν οι πόροι τους να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, γιατί αυτό εδώ δεν το εγγυόμαστε με αυτά τα αποτελέσματα. Ε, ε, ε, λοιπόν, μου είπαν ότι η Κομισιόν δεν έχει σκοπό να μιλήσει για το θέμα αυτό, άρα θα δώσουμε το λόγο Α, θέλει κάποιος να παρέμβει τελικά. Άλλο μου είπαν εδώ, δεν ξέρω. Ποιος κύριος, ποιος θα πάρει το λόγο. Μήπως δεν κατάλαβα. Και ο Σπυρόνιο θέλει το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Πυρόνιο. Oui, euh, Καλημέρα. Πυρόνιο λέγομαι. Ασχολούμαι με τα προβλήματα Τη ε, συντήρησης της χλωρίδας και της πανίδας στην Αφρική. Εδώ και 28 χρόνια ασχολούμαι το θέμα. Το ξέρω καλά το θέμα. Αυτό που θέλω να πω, καταρχήν όσον αφορά την παρέμβαση του κ. Ταουρή, είναι ότι συμμερίζομαι απόλυτα την ανάλυση του κυρίου Ντραουρή. Θα ήθελα να πω ότι ίσως θα μπορούσαμε να προχωρήσουν πιο πέρα από αυτά που ανέφερα. Αναφέρθηκε σε είδη που απειλούνται πολύ, όπως το λοντάρι, ελέφαντες και οι γορίλες. αλλά ο κίνδυνος εξαφάνισης αυτού των ειδών ξεπερνά την απώλεια των ίδιων των ειδών αλλά υπονομεύει οικοσυστήματα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε οικολογικές αναταράξεις τεράστιες. Και όπως σωστά είπε, κάτι το οποίο θα είναι μονόδρομος. Δεν θα μπορούν να επαναρθωθούν όλα αυτά αναφέρεται η προστασία των ελεφάντων για τους ελέφαντες, για το είδος, των λονταριών και τα λοντάρια Είναι αυτό, αλλά υπονομεύεται όλο το οικοσύστημα. Και μακροχρόνια αυτό που έχει τεράστιες συνέπειες όσον αφορά τους πληθυσμούς που ζουν σε αυτά τα ενδιατήματα. Οι πληθυσμοί πιο φτωχοί ζουν εκεί. Αυτοί χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους για τη ζωή τους, για την επιβίωσή τους. Και έχω και κάποιο σχόλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σχεδόν αποκλειστικό δωρητή για την προστασία της πανίδας στην Αφρική. Δίστασα να το πω, διότι και ο Σντράουρη αμφισβήτησε πολλές χρηματοδοτήσεις. Αληθεύει όμω, Πρέπει να εξεταστούν σε διάφορα επίπεδα οι δράσεις. Σε εθνικό, τοπικό, περιφερειακό επικεντρώσαμε τις προσπάθειές μας τα τελευταία 28 χρόνια στην προστασία ε, τοποθεσιών που ε, είναι σημαντική. Είναι θέμα προγραμματισμού, διαδικασιών κλπ. έπρεπε να ακολουθήσουμε και δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε σφαιρική ε, στρατηγική. Ζήτησε ο Επίτροπος που είναι υπεύθυνο τα θέματα αυτά να μας ζητήθηκε να ετοιμάσουμε στρατηγική σφαιρική σε επίπεδο τοπικό και διεθνές. Σε συνεργασία και με το Consortium για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας του τομέα, με την Interpol, προβλέπει και στρατηγική να υποστηριχθούν δομές, όπως αυτές περιέγραψε ο κύριος Ντραουρή. Η στήριξη δεν αφορά μόνο τα χρήματα, δεν ζητούν τόσο πολύ αυτό, αλλά χρειάζεται πολιτική στήριξη επίση και διπλωματική. Ετοιμάσαμε αυτή τη στρατηγική. Είναι σε τεχνικό επίπεδο η συζήτηση. Θα ακολουθηθεί η ιεραρχική προσέγγιση και ελπίζουμε να βρούμε τη δυνατότητα, θα τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη στρατηγική. Να υπογραμμίσω και κάτι άλλο που αφορά τη διαφθορά. Πολύ συχνά θεωρήσαμε ότι οι αυτοί που πήραν τι αποφάσει θεώρησαν ότι κάναμε καλό εφαρμόζοντα εσπίζοντα κανόνε για να αποφύγουμε τη διαφθορά. Και κυρίω ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτοί οι κανόνε ευνοούν καμιά φορά, αντιθέτω, ευνοούν την διαφθορά. Παράδειγμα, σήμερα αν ήθελα να παρέμβω στο Καμερούν, να βοηθήσω τον κύριο Ντραουρί σε αυτά που κάνει, που είναι πολύ καλά. Δεν θα μπορούσα να το κάνω διότι έπρεπε να περάσω μέσω προκήρυξης διαγωνισμού, υποβολής προτάσεων. Και πιθανόν οποιοδήποτε άλλος, οποιαδήποτε άλλη δομή μπορούσε να κερδίσει τη σύμβαση. Και κάποιος φορέας που να συνδέεται με τους διεφθαρμένους. Δεν έχω δικαίωμα ε, να, παρά, να τον βοηθήσω παρά την έξοχη δουλειά που κάνει. Υπάρχουν δομές που έχουμε θεσπίσει για τη διαφάνεια, για την αποφυγή της διαφθοράς, και στο επίπεδο της διαφθοράς που ευνοεί όμως τη διαφθορά διότι υποχρεώμαστε να διανύμουμε χρήματα σε δομές για τις οποίες δεν υπάρχουν εγγύσεις. Και γιατί δεν έχουμε εγγύσεις. Διότι δεν έχουμε τα μέσα ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθούμε τι γίνεται, την όλη διεργασία. Ασχολούμε με την πανίδα και την προστασία της πανίδας 28 χρόνια, τρία άτομα είμαστε για όλο τον κόσμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε χρήματα για αποστολέ. Και μας έδειξε αυτά, μας έδειξε η διευθύντρια της Όλαφ. Και τέθη γιατί δεν πήγαμε. Γιατί δεν το πήραμε είδηση πιο πριν, απλούστατα. Διότι δεν έχω χρήματα για αποστολές να πάω επί τόπου. Δεν ανήκω σε αυτούς τους τομείς, αλλά σε άλλους τομείς ε, είναι παρόμοια τα πράγματα. Δεν μπορώ να πάω να δω τι τρέχει. Άρα θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Άρα είναι ένα πρόβλημα πόρων που διατίθενται και η μείωση των πόρων για έλεγχο των πόρων που χορηγούμε. Αυτό είναι, η μείωση των πόρων για τους ελέγχους. Ε, να πω ότι συμμεριζόμαστε 100% της ανησυχίες του κυρίου Ντραουρή. Είναι κάτι που γνωρίζουμε, το συζητήσαμε και μεταξύ μας. Είναι κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε όμως και θέλω να πω ότι είναι πήγον το ζήτημα διότι όπως είπε ο κ. Ντραουρή σε 10-15 χρόνια πολλά πράγματα, πολλά είδη θα εξαφανιστούν. Αυτό είναι κάτι ανεπανόρθωτο και Αφρικανική Ήπειρος ε, θα αλλάξει ριζικά, θα αλλάξει η εικόνα της. Αυτό είναι ο κίνδυνος, να έχουμε δραματικές συνέπειες όλων αυτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαι αρμόδιος μεταξύ άλλων για την πολυγλωσία και την διερμηνία στις δραστηριότητές μας. Για τη διερμηνία ε, απομένουν 7 λεπτά αντε 12. Αν οι διερμηνείς μας ε, έχουν την καλοσύνη να δουλέψουν άλλα 5 λεπτά. Τρία λεπτά λοιπόν έχετε ο καθένας από τους τρεις ε, ομιλητές του πάνελ για να απαντήσετε στα πολλά σχόλια. Φαντάζομαι ότι θα θέλατε μια ώρα καθένας, αλλά τρία λεπτά έχετε παρόλα αυτά στη διάθεσή σας. Κύριε Πάρτο, είστε ο πρώτος για την παρέμβαση. Έχετε τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Χάσαμε το χρόνο μας με το Αφγανιστάν. Όχι. 50% του πληθυσμού είναι κάτω από την ηλικία των 25. Κάποιοι έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, όλοι έχουν ε, ζήσει περίπου ε, τη μισή του ζωή σε δημοκρατία που δεν το είχαν. Ε, μόνο και γι' αυτά αξίζει τον κόπο η παρέμβασή μας. Ε, δεν απαντώ στη δική σας ερώτηση, ήταν άλλο, σε άλλο σχόλιο απαντώ. Στη δική σας ερώτηση, τι θα γίνει το 2014. Ένα τμήμα του προβλήματος της ε, διαφθοράς είναι το ότι εισραίουν στη χώρα τεράστια ποσά που δεν μπορούν να απορροφηθούν και να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά. Αυτό το 2014 θα αλλάξει γιατί τα χρήματα θα είναι πολύ πιο λίγα. Αυτό είναι καλά νέα. Και επίση η αποστατικοποίηση είναι πολύ καλό νέο. Υπάρχουν λοιπόν αρκετέ περιπτώσει, αρκετέ μάλλον δυνατότητε, να δράσουμε τώρα ενεργά και να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τον περίοδο μετά το 2014. ΜΜΕ. Πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα εκεί. Ήδη υπάρχουν πολλά παραδείγματα για το τι γίνεται κανεί όταν κάνει προγραμματισμό χωρί να κατανοεί το ε, πλαίσιο τη χώρα. Επίση, επένδυση στην έρευνα ε, ακτιβιστικές δράσεις ε, δεν μπορούμε να τους, ε, να τους ε, στα, να σταματήσουμε την υποστήριξή μας. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που δεν εξάρτησατε το χρόνο σας. Ο κύριος Ντρόντ έχει τώρα το λόγο. Αυτό το ευχολόγιο που ζητήσατε, πιο αυστηρέ ποινές θα ήταν στο νούμερο 1 για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλλον το νούμερο 2 θα ήταν εποπτικό σύστημα ετήσιων εκθέσεων, γενικό σύστημα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, ώστε να υπάρχει εποπτεία για να μπορέσει να υπάρξει πίεση. Και τρίτο, πιο έξυπνες αποφάσεις χρηματοδότησης. Υπάρχουν πολλά εργαλεία της κοινωνίας των πολιτών που έχουν προετοιμαστεί ακριβώς γι' αυτό. Ε, η αιρεσιμότητα τώρα που αναφέρατε είναι ένας από τους τρόπους που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Αλλά επίσης υπάρχει και το Governance Investment Manual που λέει ότι για κάθε ε, επένδυση σε κάθε τομέα υπάρχει ένα κομμάτι των χρηματοδοτήσεων που θα χρηματοδοτεί συγκεκριμένα ε, projects που αυξάνουν την λογοδοσία και τη διαφάνεια σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα. Οπότε έχουμε ε, μια διαφορετική στάση απέναντι σε, αυτά τα project και έχουμε μια δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερης λογοδοσίας και διαφάνειας μέσα από τα ίδια τα project. Εγώ ε, έρχομαι ως ε, εκπρόσωπος της ε, κυβέρνησης του Καμερούν από την σχετική διάσκεψη που ήταν πραγματικά πολύ απογοητευτική για την σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της διαφοράς από την διάσκεψη ΣΑΙΤΕΣ. δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Για την βοήθεια τώρα στους κυνηγού. δεν αμφισβητώ τα, ότι τα παραδείγματα που έχουμε εμείς είναι παραδείγματα όπου οι κυνηγοί σαφάρι ε, ξέπλαιναν πολλά χρήματα, αλλά ξέρουν και πώς μπορούν να, φέρ, να στείλουν χρήματα πίσω στους τόπους αυτούς της ε, διατήρησης ε, ή τους οικοτόπους. Βέβαια υπάρχουν δυνατότητες να βρεθούν οι ροές αυτών των χρημάτων. Τώρα για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που αναφέρατε. Μη κυβερνητικέ οργανώσεις και διαφθορά. Αυτό το θέμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ε, ερευνήσαμε πάρα πολύ το τι γίνεται με τις ΜΚΟ. Υπάρχουν πολλοί ε, κανονισμοί που μπορούμε να προωθήσουμε για τις ΜΚΟ για να αυξήσουμε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Έχουμε δει μεγάλα θέματα διαφθοράς εντός των ΜΚΟ που είναι ακόμη πιο λίγη η λογοδοσία τους από τις κυβερνήσεις των, του αναπτυσσόμενου κόσμου. Και επίσης δόθηκε μια πολύ σαφής εικόνα για το τι γίνεται με το περιβάλλον. Αλλά αυτό είναι ένας από τους τομείς. Πρέπει να βάλουμε την, ε, τον αγώνα της ε, ε, για την αντιμετώπιση διαφθορά, στον πυρήνα των προσπαθειών μας, των ε, ε, δαπανών μας, για να αλλάξουμε γενικώ συμπεριφορά και το πώ χρησιμοποιούμε τα χρήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. κύριε κυρία έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω ουσιαστικά. Η μία φορά τη συζήτηση ΕΠΟ για αύριο δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Ε, αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το διασυνοριακό έγκλημα με διασυνοριακούς ε, ανακριτές και ελεγκτές. Θα πρέπει κάτω από την ίδια μπρέλα να βάλουμε όλους τους εμπειρογνώμονες από τους διάφορους τομείς. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Νίτον Ντάν, συμφωνώ, όπως είπατε, ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτή την κατεύθυνση βέβαια τα κράτη-μέλη και η Όλαφ. Πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Αν και μου φαίνεται κάποιες φορές σαν να πυροβολούμε με νερομπίστολα, τέλος πάντων. Ένας φορέας που αναφέρατε, ε, αυτό το δικαστήριο, αυτό το ζώο το ευρωπαϊκό, θα ήταν κάτι θετικό και θα μας ε, βοηθούσε να προστατεύσουμε τα θύματα ή τη ε, φορολογούμενους ή τα, τους ανθρώπους και τα ζώα που είναι θύματα. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα της κυρίας, συγγνώμη δεν διαβάζω από τόσο μακριά το όνομά σας. Μπορεί να είναι θέμα παρακολούθησης και ελέγχου. Το θέμα είναι ποιος υποτίθεται ότι αναλαμβάνει αυτό το έργο. Μπορεί η Κομισιόν όταν ε, δίνει κάποια χρήματα να ακολουθεί ε, το ίχνος τους σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι μια διαφορετική υπόθεση η ευθύνη που έχει η Κομισιόν μετά τη χρηματοδότηση. Βέβαια θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τις χώρες στις οποίες ε, δίνουμε, εκταμιεύουμε πόρους, ώστε να αναλάβουν την ευθύνη να οικειοποιηθούν τις διαδικασίες αυτές. Τι μπορούμε να κάνουμε θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου. Αλλά η διαφθορά που γίνεται από τους ε, υπαλλήλους ε, είναι πολύπλοκη, δύσκολο να ανοιχνευτεί πολλές φορές. στη Γερμανία που ήταν να ανοίξει τον αεροδρόμιο βρήκαν προβλήματα και βλέπετε ότι ακόμη και σε προηγμένες χώρες ε, δημιουργούνται τέτοια θέματα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της ε, συνεδρίας αυτής που ήταν ε, συναρπαστική. Αν μου επιτρέπετε, ένα τελευταίο σχόλιο, έτσι μια απόχρωση να δώσω σε αυτά που είπε ο κύριος ο βετεράνος στον τομέα του. Εδώ και κάποιους μήνες αυτό το οποίο έχουμε σε όλες τις χώρες που γίνονται προγράμματα, έργα, έχουμε μία πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα πρέσβη και έχουμε και προσωπικό. Αυτό το προσωπικό πρέπει και αυτό να αναλάβει ευθύνες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πηγαίνει στην Κεντρική Αφρική ο κύριος Πυρώνιο γιατί στην Κεντρική Αφρική, σε κάθε μία τη χώρες Κεντρική Αφρική υπάρχει πρεσβεία, υπάρχει προσωπικό που θα έπρεπε, θα έπρεπε να έχει ευθύνη να παρακολουθεί τα έργα, τα project τα οποία υλοποιούνται εκεί και να παρακολουθεί την κατάσταση, όπως πολύ καλά είπε ο συνάδελφός μας, για να μην έχουμε αυτή την καταστροφή που είδαμε με το ε, νοσοκομείο που έγινε τελικά φαρσοκομωδία μετά από τρία χρόνια. Αυτά που μας είπε ο κ. Σπυρών είναι πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα και εμεί από πλευρά Κοινοβουλίου θα επιμείνουμε Αυτή οι πρέσβη, που δεν είναι πρέσβης της Κομισιόν, εκπρόσωποι τη Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πρέσβη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και του Κοινοβουλίου. Πρέπει να έχουμε τον έλεγχο, Εμεί να έχουμε τον έλεγχο, ότι το προσωπικό αυτό παρακολουθεί, επιβλέπει στην πράξη τα έργα τα οποία υλοποιούνται στην επικράτηση χώρα στην οποία βρίσκονται και τα οποία αυτά έργα χρηματοδοτούνται με πόρους των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Νομίζω ότι πραγματικά είναι μία ε, κλίση στην τάξη μας. Ε, μας καλούν στην τάξη όλοι με αυτά που μας λένε εδώ αυτή σε αυτή την ακρόαση και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, όλοι μας μας ανακαλούν στην τάξη για να μην έχουμε καταστροφές σαν αυτές που είδαμε στις οθόνες. Ευχαριστώ τους φίλους, τις φίλες, όλους όσους παρακολούθησαν την ε, σημερινή μας ακρόαση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους βουλευτές, οι οποίοι όλοι μας φαντάζομαι μάθαμε πολλά. Μας ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ακρόαση και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες και το προσωπικό της Επιτροπής Ανάπτυξης που διευκόλυνε τόσο πολύ τη δουλειά μας. Κλείνει η συνεδρίαση αυτή και θα τα πούμε το μεσημέρι εμείς, ε, γιατί έχουμε την ε, πολύ σημαντική συνεδρίαση του απογεύματος με ψηφοφορίες στην Επιτροπή